Καλημέρα σας, κυρία Ξεκι... Ξεκινάμε πάλι με την ημερήσια διάταξη που αφήσαμε χτες. Είμαστε στο σημείο της ψηφοφορίας και επειδή θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά θα ήθελα να δοκιμάσουμε, αν συμφωνείτε κι εσείς, Έχετε όλοι τις κάρτες σας. Α, λείπει μια κάρτα. Η κυρία Γκρέσλε. Ξέχασα την κάρτα της κυρία Γκρέσλε. Ξεκινάμε λοιπόν. Ψηφίστε για να κάνουμε μια δοκιμή του συστήματος. Ελέγχουμε λοιπόν το ηλεκτρονικό σύστημα. Okay. Äh, komme ich äh, zur Abstimmung. Και τώρα μπορούμε να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Έχουμε τον κανονισμό για την ε, Όλαφ. Έχουμε ουσιαστικά την πρώτη ψηφοφορία, η συγγήτρια η κυρία Γκρέσλε, πρόκειται για το 1073-1999. Η συγγήτρια έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω ότι σήμερα ψηφίζουμε το κείμενο του Συμβουλίου. Γιατί έχουμε πει στο Συμβούλιο ότι θα υποβάλει τροπολογίες. Η ομάδα μου όμως, και πιστεύω ότι και άλλες ομάδες θα συμφωνήσουν και θα εκφραστούν έτσι στην Ολομέλεια. Θεωρούμε ότι ο έλεγχος προς την Όλαφ χρειάζεται ενδυνάμωση. Εξού και θεωρούμε ότι θα πρέπει κάποιες από τις προτάσεις να αναδιατυπωθούν και να γίνουν πιο συγκεκριμένες. Πρόκειται λοιπόν για τρεις τροπολογίες. Θα προσπαθήσουμε να τις συγκεντρώσουμε με τεχνικό τρόπο έτσι ώστε να παρουσιάσουμε νέα ε, κείμενα. Υπάρχει και μία επιπλέον τροπολογία η οποία θα υποβληθεί που αφορά το θέμα της αμφισβήτησης μίας ε, έκθεσης ε, της Όλαφ ενώπιον των δικαστικών αρχών. Αυτό σήμερα δεν επιτρέπεται. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα αμφισβήτησης από την Όλαφ ενώπιον των δικαστικών αρχών και είναι υποχρεωτικό σήμερα να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτή τη δυνατότητα, να μπορεί δηλαδή κανείς να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να αμφισβητήσει μία έκθεση της Όλαφ. Η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών είναι η επόμενη εβδομάδα. Σας παρακαλώ πολύ λοιπόν να δεχτείτε την πρότασή μου. Θεωρώ πραγματικά ότι υπάρχουν σημεία του κειμένου τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαριστούν, να αποσαφηνηθούν περισσότερο, να γίνουν πιο συγκεκριμένα και θεωρώ επίσης ότι σήμερα δεν πρέπει να ψηφίσουμε διότι την επόμενη... θα ψηφίσουμε δηλαδή για τις ε, σημερινές προτάσεις, αλλά την επόμενη εβδομάδα να ξέρετε ότι θα υποβληθούν και άλλες προτάσεις. Ωραία, πρόεδρος. Μπορούμε να κάνουμε καταρχήν την ε, πρώτη ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 16 ναι. Κανείς κατά, κανείς δεν απέχει. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία, που είναι η έγκριση του σχεδίου γνωμοδότησης. Προϋπολογισμός 2014, ο Γιάννης Γκάιερ είναι ο εισηγητής. Εδώ έχουμε διάφορες ψηφοφορίες ξεχωριστές για την παράγραφο 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4, τροπολογία 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 7 υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 7, λέει ο πρόεδρος. Check is... Τέλος ε, της ε, ψηφοφορίας. 10 υπέρ, 6 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. 6. Τροπολογία 6. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 7. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Παράγραφος 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δέλτα. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το ψήφισμα συνολικά ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. 16 υπέρ. Μία ψήφος κατά μία αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν το ψήφισμα και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ψηφοφορία που είναι η έκθεση Ντελάνγκε προς μια αποτελεσματική και οικονομική αποδοτική διερμηνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 4. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Εννέα. Όχι. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται αυτή η τροπολογία. Δεν μπορέσατε να ψηφίσετε. Δουλεύει το σύστημα, δουλεύει το μηχανημά σας. Ωραία, επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Ξαναψηφίζουμε την τροπολογία 4, αρχή της ψηφοφορίας. open. Everybody voted? No? Okay. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Η κυρία Γκρέσλε δεν έχει όμως κάρτα. Είστε κατά. 10 υπέρ 10 κατά. Δεν περνάει αυτή η τροπολογία. Κρίμα. 5. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία, τροπολογία 6. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Όχι. Αρχή της ψηφοφορίας. Τέλος. Κυρία Γκρέσλε, υπέρ. 11 υπέρ 8 κατά. 7. Τροπολογία 7. Υπέρ υπέρ της 7, κατά της 7, αποχές, απορρίπτεται η 7. Ρούμπικ, προφορική τροπολογία του κυρίου Ρούμπικ, υπέρ. Η εισηγήτρια. Για να... να είμαστε απολύτως ακριβείς. Ε. Θα ήθελα στο κείμενο αυτή της προφορικής τροπολογίας του κυρίου Ρούμπιχ να προσθέσω κάτι. Έχετε το κείμενο, επιμένει ότι κτλ. κτλ. Μετά το επιμένει ότι θα ήθελα να προσθέσω Σεβόμενη τις αποφάσεις ε, του Προεδρείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ε, πολυφωνία και τον σεβασμό των, ε, του λεσκού καθεστώτος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά να προσθέσουμε την συνέχεια του, της τροπολογίας του κυρίου Ρούμπιχ έτσι όπως τη δέχεται μπροστά σας. Συμφωνείτε όλοι με αυτή την αποσαφήνιση της συγκητρίας, αντιτίθεται κανείς, όχι. Λέει ο πρόεδρος, πως μπορούμε να ψηφίσουμε επί της προφορικής τροπολογίας με την προσθήκη του συγκητρίας. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά. Αποχέ. εγκρίνεται. 11 υπέρ, κατά έλεγχος. Τροπολογία 10. Η 11 λέει ήταν ο πρόεδρος, μάλιστα η 11. Ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται. Ε, ψήφισαν όλοι, πέρας. 11 υπέρ, 8 κατά, επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά. Αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Eh, Τροπολογία 12. Ευχαριστώ. Everybody voted. Vote is closed. It is uh, rejected. Απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη 13. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Α, να ελέγξουμε την 3. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για την τροπολογία 3. κυρία Γκρέσλε. Είστε υπέρ ή κατά. Ωραία. 12 υπέρ, 9 κατά. Απορρίπτεται. Α, συγγνώμη. Απορρίπτεται, άρα 12 κατά, 9 υπέρ. Ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου. Ψηφίζετε όλοι. Πέρα τη ηλεκτρονική ψηφοφορία. 20 υπέρ 0 κατά συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τους εισηγητές, τις εισηγήτριες, τα μέλη της γραμματείας που μας βοήθησαν και νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε με την ημερήσια διάταξη. Είμαστε στο σημείο 12 και πρόκειται για την ετήσια έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας της Όλαφ, έρευνες της Όλαφ, ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης, την Όλαφ. Σήμερα θα υπάρξει ανταλλαγή απόψεων παρουσία του Γενικού Διευθυντού της Όλαφ, Τζοβάνι Κέσλερ, Γενικού Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης. Σας καλωσορίζω κύριε Κέσλερ. Μεγάλη φασαρία βέβαια εδώ στην αίθουσα. Όποιος θα ήθελε να συζητήσει μπορεί να βγει έξω από την αίθουσα. Κύριε Κέσλερ, καλωσορίσατε στην τελευταία συνεδρίαση. Δεν μπορέσαμε να ανταλλάξουμε απόψεις μαζί σας, διότι είχαμε θέμα χρόνου, περιμέναμε και κάποιες μεταφράσεις κειμένων. Σκοπός μας είναι να ξεκινήσουμε ένα διάλογο μαζί σας. Ε, φαντάζομαι ότι όλοι οι παρόντες θα είναι πολύ πειθαρχημένοι Εχθές στη συνάντηση των συντονιστών συμφωνήσαμε ότι επιθυμούμε μία διαδικασία που ισχύει για τις ακροάσεις των επιτρόπων, δηλαδή εμείς θα κάνουμε σύντομες ερωτήσεις, περιορισμένου χρόνου αν θέλετε, έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι να κάνουν ερωτήσεις και να υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Ένα λεπτό λοιπόν διάρκεια των ερωτήσεων. Κύριε Κέσλερ, θα σας ζητήσω επίσης να απαντήσετε κάθε φορά μέσα σε δύο λεπτά. Έτσι ώστε σήμερα το πρωί να μπορέσουν όλοι οι συνάδελφοι να θέσουν τις ερωτήσεις που επιθυμούν. Υπάρχει το ερωτηματολόγιο το οποίο σας έχουμε στείλει, το οποίο έχουμε απευθύνει στην Επιτροπή Εποπτείας της Όλαφ και στην ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δυστυχώς, δυστυχώς διαπιστώσαμε ότι το 40% των ερωτήσεων δεν απαντήθηκαν, δεν μπόρεσαν να απαντηθούν μας είπαν διότι πρόκειται για θέματα που αφορούν ε, την διαδικασία που είναι εν εξελίξη σε περιπτώσεις που εμείς είχαμε την εντύπωση ότι θα μπορούσαν να είχαν απαντηθεί οι ερωτήσεις ενώ παραδείγματο χάρη είχαν ανακοινωθεί διάφορα στοιχεία ή διάφορα τμήματα απαντήσεων ήδη στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στον τύπο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι κάτι που δημιούργησε μια δυσαρέσκεια και θα θέλαμε εδώ πραγματικά να επιστήσουμε την προσοχή σας στο θέμα της προσοχής προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Υπάρχει η υπόθεση του Επιτρόπου Ντάλι και εδώ και πολλούς μήνες περιμένουμε κάποιες συγκεκριμένες απαντήσεις. Τέλος Μαΐου η συνδιάσκεψη των Προέδρων έθιξε το θέμα αυτό από κοινού με την ε, υπόθεση της ε, ετήσιας έκθεσης της Επιτροπής Εποπτείας της Όλαφ και γι' αυτό και εμείς ε, θέλουμε να επανέλθει το θέμα αυτό δεν δεχόμαστε να στέλνουμε, να απευθύνουμε ερωτήσεις οι οποίες μένουν αναπάντητες, ενώ την ίδια ώρα υπάρχουν τοποθετήσεις και δηλώσεις στον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εμείς ε, ερμηνεύουμε αυτήν την στάση με έναν τρόπο που πραγματικά μας ε, δυσαρεστεί ε, και τα εισαγωγικά μου σχόλια είναι ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να συνεχίσει αυτή η αντιμετώπιση. Υπάρχουν λοιπόν πολλές ερωτήσεις που θα σας ε, τεθούν από τα διάφορα μέλη της ε, Επιτροπής. Κύριε Κέσλερ, ήσασταν παρόν και στην τελευταία μας συνεδρίαση, δεν προλάβαμε όμως να κάνουμε τις ερωτήσεις ε, που θέλαμε. Θα ζητήσω λοιπόν καταρχήν... Α, ο κύριος Κάλβιν έχει ένα διαδικαστικό. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί δεν ε, ήμουν ε, στους συντονιστές ούτε ο αναπληρωτής μου. Και ο συνάδελφος Γκάρντ δεν μπορεί να είναι ούτε σήμερα. Εν πάση περιπτώσει, Βεβαίως ε, στηρίζουμε απολύτως την διαδικασία την οποία προτείνεται και πραγματικά πρέπει να έχουμε χρόνο για να απαντήσει ο, ο, ο κύριος Κέσλερ όσο γίνεται σε περισσότερες ερωτήσεις γιατί ξέρουμε τι έγινε την προηγούμενη συνεδρίαση. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε στον Γενικό Γραμματέα ίσως πέντε λεπτά για να κάνει ίσως κάποια πρώτη τοποθέτηση. Κοιτάξτε, εμείς δεν είμαστε διερευνητική επιτροπή. Ίσως σε μια κανονική συζήτηση μπορεί κανείς ε, να ε, περιορίσει την συζήτηση στα πέντε λεπτά. Ναι, αυτό είναι θέμα διαδικασίας. Κυρία Κρέσλε και οι άλλοι συντονιστέ, τι έχετε να πείτε. Ο Γενικός Διευθυντής στην τελευταία συνεδρίαση μίλησε επί 45 λεπτά. Δεν μπορούμε να πούμε ότι του περιορίσαμε το χρόνο Λίας. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να απαντήσει και στις ερωτήσεις μας. Μίλησε επί 45 λεπτά. Δεν είμαστε υπέρ λοιπόν να του ξαναδοθεί ο λόγος. Ποιος άλλο θα ήθελε να πάρει το λόγο ή θα ψηφίσουμε. Ο κύριος Στάς. Θα ήθελα να συμφωνήσω με την κυρία Γκρέσλερ. Κοιτάξτε, ούτως ή άλλως έχουμε και ένα έγγραφο εννέα σελίδων περίπου όπου ε, αναφέρονται όλα αυτά τα οποία ε, είπε η κυρία Κρέσλερ. 45 λεπτά μίλησε ο κύριος Κέσλερ την προηγούμενη φορά. Ε, ξέρουμε πολύ καλά τι είπε και γνωρίζει ότι το Κοινοβούλιο έχει ε, πολλές ανησυχίες όσον αφορά κάποιες κατηγορίες οι οποίες ακούστηκαν. Πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε τα ερωτήματά μας. Λοιπόν, υπάρχει μια συγκεκριμένη πρόταση του κυρίου Κάλφιν να ψηφίσουμε. Ποιο είναι υπέρ του να δοθεί λίγο χρόνο ομιλία στο Γενικό Διευθυντή τη Όλαφ. Σηκώσε το χέρι. Υπέρ. Άντε, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Ποιο είναι υπέρ του να δώσουμε καταρχήν το λόγο στον ε, Γενικό Διευθυντή της Όλαφ, να κάνει κάποια εισαγωγικά σχόλια. Ψηφίζουμε. Ε, okay. Now. Ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Τέλος. Ξαναψηφίζουμε. Check is open. Αρχή της ψηφοφορίας. Οχτώ υπέρ, Κυρία Γκρέσλε, ψηφίσατε. 8 υπέρ, 8 κατά. Απορρίπτεται. Και μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στη διαδικασία των ερωτήσεων και απαντήσεων. Έχουμε τους επικεφαλείς, συγγνώμη, τους συντονιστές των πολιτικών ε, ομάδων και παρακαλώ πολύ τη γραμματεία να προσέχει το χρόνο. Η κυρία Γκρέσλε, το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Γενικέ Διευθυντά, σας ευχαριστώ που δέχεστε αυτή την ανταλλαγή στην ZDF στις 3 Απριλίου είπατε ότι σε μια συνέντευξη ότι ουσιαστικά οι παρακολουθήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων έγινε χωρίς να είναι γνωστή αυτή η διαδικασία. Απ' την άλλη είπατε ότι είναι μια νόμιμη και κανονική διαδικασία. Αυτό που ξεχάσατε να πείτε είναι ότι από τη στιγμή που ένας συνομιλητής γνωρίζει την ύπαρξη της παρακολούθησης, της διαδικασίας παρακολούθησης και ο άλλος όχι, δεν είναι νόμιμη. Και αυτό βεβαίως και βάσει του ποινικού κώδικα του Βελγίου αλλά και βάσει της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Πρόκειται για διαδικασίες που δεν είναι νόμιμες και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να τις θεωρήσουμε αποδεκτές. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Τηρήσατε και το χρόνο ομιλία σας και κάνατε μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ο κύριος Κέσλερ έχει το λόγο για την απάντησή του. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, 15 δευτερόλεπτα κυρία ε, Κρέσελ για να σας ε, ζητήσω την ευγένειά σας και ε, να κάνω κάποιες σκέψεις και κάποιες επεξηγήσεις ε, τις οποίες ε, έχω γράψει. Δεν ήξερα πώς θα ε, λάβει χώρα αυτή η συνεδρίαση και έγραψα κάποιες σκέψεις τις οποίες θεώρησα χρήσιμες για το Κοινοβούλιο. Θα σας την μοιράσω αν μου το επιτρέπετε τις σημειώσεις αυτές στο τέλος της συνεδρίασης. Και βεβαίως τώρα θα απαντήσω στις ερωτήσεις. Αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο σας υποβάλλω. Πρόεδρος, να σας διακόψω. Και βεβαίως δεν μετράει αυτός ο χρόνος. Ε, τα έχουμε ήδη μοιράσει τα γραπτά σας σχόλια, τα έχουν ήδη τα μέλη. Ωραία, πολύ ωραία λέει ο κύριος Κέσλερ, πολύ ωραία, δεν με είχαν πληροφορήσει γι' αυτό. Ε, ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ε, καλό θα ήταν λοιπόν να απαντήσετε και τη συγκεκριμένη ερώτηση τώρα. Ναι, φυσικά λέει ο κύριος Κέσλερ. Πρώτα απ' όλα, το, ζήτημα της ε, συστηματικότητας ε, ε, βεβαίως δεν ισχύει. Εγώ το αρνούμαι. Δεν είναι κάτι συστηματικό. Αυτό που συνέβη σε αυτή τη διερεύνηση της συγκεκριμένη υπόθεσης είναι ότι δύο φορές τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μεταξύ ιδιωτών παρακολουθήθηκαν στην πρώτη περίπτωση πριν την έναρξη της διαρευνητικής διαδικασίας, δεν ξέραμε δηλαδή καθόλου ως όλα ότι αυτό συνέβαινε, ούτε συμμετείχαμε με οποιοδήποτε τρόπο, ε, γιατί ξέρετε ότι ένας ιδιώτης μπορεί να καταγράψει μια τηλεφωνική συνδιάλεξη που έχει με έναν άλλο ιδιώτη. Η καταγραφή αυτής της τηλεφωνικής συνδιάλεξης εκ των υστέρων εδόθη στην Όλαφ ως στοιχείο αποδεικτικό στα πλαίσια της διερευνητικής διαδικασίας. Υπήρξε άλλη μία περίπτωση παρακολούθησης, δηλαδή το ίδιο άτομο έκανε το ίδιο πράγμα δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια της διερευνητικής διαδικασίας τη, ε, ε, παρουσία των ε, ερευνητών της Όλαφ. Ε, στα πλαίσια της ε, διαδικασίας που έλαβε χώρα στην Επιτροπή Εποπτείας και την οποία συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Δεν υπάρχει καμία παραβίαση εδώ του βελγικού νόμου και επίσης ε, δεν υπάρχει και καμία παραβίαση οποιοδήποτε ανθρωπίνου θεμελιώδους δικαιώματος. Βεβαίως θα μπορούσε και θα συζητηθεί ενδεχομένως ε, στα δικαστήρια η υπόθεση αυτή εάν εγείρει ζήτημα ε, ο ενδιαφερόμενος. Όμως, οτιδήποτε συνέβη αφενός δεν είναι συστηματικό, αφετέρου είναι πλήρως νόμιμο. vielen Dank, äh, dass die Zeit... Ευχαριστώ πολύ. Τηρήσατε και εσείς το χρόνο ομιλία σας. Η κυρία Γκρέσλη για ένα λεπτό. Μα αυτό είναι το περίεργο. Εδώ πρόκειται για πλήρη και προφανή παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Και ακούω κάποιον πίσω μου να λέει ότι είναι κάτι το νόμιμο. Υπάρχει η ανάλυση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου και θα ήθελα να μας αποσταλεί. Έχει ανακοινωθεί ότι υπάρχει, ότι έχει γίνει αυτή η νομική ανάλυση, γιατί δεν μας έχει ακόμα δοθεί. Πρέπει επίσης να προσθέσω ότι η πρώτη τηλεφωνική συνδιάλεξη, χωρίς δηλαδή τη συμμετοχή της ε, Όλαφ, ε, ε, χρησιμοποιήθηκε στην διαρεύνηση της Όλαφ ως στοιχείο αποδεικτικό. Το δεύτερο τηλεφώνημα ούτε μεταγράφηκε, ούτε χρησιμοποιήθηκε με οποιοδήποτε τρόπο ως ε, μαρτυρία ή ως αποδεικτικό στοιχείο ε, στην ε, διαρευνητική διαδικασία και επομένως δεν προκύπτει καμία παραβίαση οποιοδήποτε δικαιώματος. Αναφέρεται και στην αναφορά μας, είμαστε απόλυτα διαφανείς, δεν συνέβη κάτι τέτοιο, δεν χρησιμοποιήθηκε και επομένως το στοιχείο αυτό και επομένως δεν είχε καμία επίπτωση στη διαδικασία. Ευχαριστώ. Äh, Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάλφιν ε, από τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξεκολουθώ να πιστεύω ότι η Επιτροπή μας δεν είναι αυτή που θα πρέπει να καθορίσει τι είναι νόμιμο, τι δεν είναι και τι θα πρέπει να διερευνηθεί ή όχι. Πραγματικά ε, νιώθω κάποια μηχανία ε, με τον τρόπο με τον οποίο ξεκινήσαμε τη σημερινή μας ε, συνεδρίαση. Τα δύο λεπτά λοιπόν της ερώτησής μου θα τα παραχωρήσω στον κύριο Κέσλερ για να θέσει το πλαίσιο γιατί έτσι νομίζω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε. Κύριε Κέσλερ, θα σας παρακαλέσω ε, να κάνετε έτσι μια σύντομη παρουσίαση στο δίληπτο που θα είχα εγώ στη διάθεσή μου. Κέσλερ, σας ευχαριστώ πολύ. Ακούστε, ευρώ, εδώ βρισκόμαστε διότι και νομίζω ότι θα ήταν ίσως ενδιαφέρον για όλα τα με Κάποιος γελάει, δεν ξέρω, τέλος πάντων. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον, αλλά τέλος πάντων. Πέρυσι το Μάιο, είμαστε λοιπόν εδώ γιατί πέρυσι το Μάιο λάβαμε επίσημη καταγγελία, ανακοίνωση από την Κομισιόν με, για μια σοβαρή, ε, ένα σοβαρό ισχυρισμό ότι η νομοθετική διαδικασία της Κομισιόν σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση της οδηγίας για τα καπνά ενδεχομένως επηρεάζεται ε, και με κάποιο χρηματικό ποσό και τέλος πάντων φάνηκε να μην είναι ε, οι διαδικασίες σωστές, να πωλείται κατά κάποιο τρόπο αν θέλετε η νομοθεσία. Και φυσικά αυτό που καταλαβαίνει ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο και για την αξιοπιστία και για τη φήμη της Κομισιόν και γενικότερα της Ένωσης. Η Όλαφ δεσμεύεται, έχει το καθήκον αυτό και έτσι ξεκίνησε γρήγορα την έρευνα όπως έπρεπε να πράξει Σεβόμενη απόλυτα την εμπιστευτικότητα του ζητήματος, το απόρριτο του θέματος και η έρευνα που δεν είχε καμία απολύτως εξωτερική ε, επιρροή ή πίεση, ήταν πλήρως ανεξάρτητη, ήταν ε, μια επαγγελματική και πρέπει να σας πω ανοιχτά ότι είμαι υπερήφανο για τον τρόπο με τον οποίο οι ερευνητέ τη υπηρεσία μου έφεραν σε πέρα σε αυτή την αποστολή. Είχαμε λοιπόν στο τέλος όλα τα στοιχεία στη διάθεσή μας, τα στοιχεία που είχαμε συλλέξει με την έκθεση, στείλαμε την έκθεση, πάντα σύμφωνα με τον κανονισμό, με το νομοθετικό πλαίσιο τη Όλαφ, στα πολιτικά θεσμικά όργανα, ουσιαστικά δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το οικείο όργανο το οποίο έπρεπε να λάβει υπόψη την έκθεση και να συναγάγει τα συμπεράσματά της. Η Κομισιόν πράγματι έλαβε την πολιτική, τις πολιτικές αποφάσεις, ε, κατέληξε στα πολιτικά συμπεράσματα. Επίσης το διαβιβάσαμε και στις αρμόδιες δικαστικές αρχές προς εξέταση το έγγραφο αυτό και ενδεχομένως ε, να ε, χρειαστεί να ληφθεί απόφαση σύμφωνα με το ε, ποινικό δίκαιο. Αυτό που βλέπουμε να συνέβη είναι ότι άλλοι φορείς έλαβαν την πολιτική απόφαση στην Μάλτα έγινε και η δικαστική διαδικασία και καταδικάστηκε ένας άνθρωπος και υπάρχει συνέχεια της διαδικασίας στη Μάλτα. Άρα αυτό που συνέβη εδώ νομίζω είναι κάτι πολύ σημαντικό. Ήτι τα θεσμικά όργανα απέναντι σε αυτή την εξωτερική απειλή νομίζω ότι αντέδρασαν κατά τον βέλτιστο δυνατό τρόπο. Äh, Ευχαριστώ πολύ και μπορούμε να περάσουμε στον επόμενο συντονιστή. Ένα λεπτό έχετε. Θα είμαι σύντομος. Κύριε Γενική Διευθυντά, μετά την έρευνα και όλα όσα συνέβησαν βέβαια με την υπόθεση Νταλή, το κοινοβούλιο μας αλλά και άλλοι οργανισμοί, άλλοι φορείς ε, ε, επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον. Ε, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ξαναρχίζατε από την αρχή θα κάνετε κάτι διαφορετικό. Κέσλερ, ένα λεπτό. Τι να πω σε ένα λεπτό. Λοιπόν, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δεν θα έκανα τίποτε διαφορετικό. Πάντα βέβαια μπορεί κάποιος να διδαχθεί από τις πράξεις του. Αλλά αυτά που τα οποία συνέβησαν στη συνέχεια αυτή η εκστρατεία, αυτή η ψευδής ισχυρισμή, τα κατασκευασμένα έγγραφα, αυτές οι μερικές ε, διαρροές ε, που στρέφονταν κατά της έρευνας της όλα, θα έλεγα και κατά της ανεξαρτησίας της, αν αυτό θα με επηρέαζε και θα έκανα κάτι διαφορετικό την επόμενη φορά. Θα κατέστρεφα την ανεξαρτησία της όλα, θα το έκανα, άρα δεν θα το έκανα. Θα συνέχισα λοιπόν με τον ίδιο τρόπο και έτσι θα συνεχίσουμε να διεξάγουμε τις έρευνές μας με τον ίδιο επαγγελματισμό, την ίδια ανεξαρτησία. Ακόμη και αν κάποιες ε, έρευνες ε, ε, ενδέχεται να οδηγήσουν σε κάποιο κίνδυνο για μας, δηλαδή να δεχθούμε πολιτικού χαρακτήρα επιθέσεις. Ευχαριστώ. Vielen Dank. Dann kommt als nächstes die alde äh, η άλλη του ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου έχει κάποια σχέση, έχει να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η όλα ε, τα στοιχεία και τα γεγονότα μετά την ε, διερεύνηση και κυρίως το γεγονός της διαρροής προς τον τύπο. Αυτό που συνέβη είναι ότι ο τύπος δεν είχε πλήρη πληροφόρηση ο ε, κατηγορούμενος επίτροπος δεν είχε πρόσβαση σε όλη την πληροφόρηση και επομένως πώς μπορείτε να πάτε στον τύπο χωρίς να έχει ο κατηγορούμενος τη δυνατότητα να υπερασπίσει τον εαυτό του. Συζητήσατε το θέμα αυτό με τον πρόεδρο ε, της ε, Κομισιόν, την πρόθεσή σας, δηλαδή το γραφείο του, την πρόθεσή σας να πληροφορήσετε τον τύπο και γνωρίζοντας ότι ο κατηγορούμενος δεν ήταν σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Απάντηση. Δύο λεπτά κύριε Κέσλερ, πάντα καλό. Απάντηση. Το κατά πόσον συζήτησα με τον τύπο και τι ακριβώς ε, διέρευσε στον τύπο. Εν τω μεταξύ είχε υπάρξει η παρέτηση του ε, του Επιτρόπου. Άρα αυτό ήταν ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός. Εμείς δεν είπαμε τίποτα. Δεν είπαμε τίποτα για την υπόθεση ούτε μετά το τέλος. Υπήρξαν και άλλες ε, περιπτώσεις ε, μεγάλων ερευνών, αλλά εμείς δεν τις αναφέραμε ποτέ στον τύπο. Όμως, όμως υπήρξε αυτό το μεγάλο νέο της παρέτησης του Επιτρόπου, που έγινε πρωτοσέλιδο παντού. Ήταν, είναι λοιπόν αφελές να ε, θεωρεί κανείς ε, ότι δεν θα ερχόταν κανένας εκπρόσωπος του τύπου σε επαφή μαζί μας. Για λόγους λοιπόν οργανωτικούς θεωρήσαμε ότι ήταν καλύτερο και πλέον διαφανές και πλέον κομψό αν θέλετε στο τέλος τις ε, συνήθους ε, ε, συνέντευξης τύπου που δίνει η Κομισιόν και αυτό είναι μια οργανωτική διαδικασία να πούμε κάποια πράγματα γιατί ήταν πιο εύκολο να το κάνουμε έτσι παρά να απαντάμε κάθε μισή ώρα σε κάποιες ερωτήσεις που υπεβάλλονται στην Όλαφ. Δεύτερον, αν θεωρώ ότι αυτό είναι δίκαιο απέναντι στον κατηγορούμενο επίτροπο. Ναι, βεβαίως. Διότι εμείς, και όχι μόνο σε αυτήν την συνέντευξη τύπου, την μοναδική άλλωστη, την οποία κάναμε μετά από την παρέτηση του Επιτρόπου λόγω του σάλου που είχε δημιουργηθεί, αλλά και στη δική σας Επιτροπή, α όχι όχι, στην Επιτροπή Κόντ, ναι, στο, ε, στο Στρασβούργο, είχε υποθεί ότι θα ήταν άδικο να σας έδινα την έκθεση και να σας παρουσίαζα όλα τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είχαμε σε σχέση με τον Επίτροπο γιατί είπαμε ότι θα πρέπει να γίνει σεβαστός ο κανονισμός και η διαδικασία. Αυτό που είπαμε λοιπόν στην λόγω συνέντευξη τύπου ε, είναι ότι είχαμε κάποια στοιχεία τα οποία δεν οδηγούσαν ε, σε απαγγελία κατηγορίας είπαμε ότι υπήρχαν υπόνοιες και ε, ενδεικτικά στοιχεία, ε, χρώσες ενδείξεις εν πάση περιπτώσει για ενδεχόμενη κατηγορία κατά του Επιτρόπου. Και αυτό που κάναμε όλους αυτούς τους μήνες ήταν το ε, ακριβώς το αντίθετο. Όλες αυτές οι κατασκευασμένες κατηγορίες απέναντι μας ε, κατασκευάστηκαν πρώτα και διέρευσαν αργότερα. Ε, έτσι ώστε να μας οδηγήσει σε, μια, ε, σε ένα είδος δημόσιας δίκης ας πούμε. Κοιτάξτε, κύριε Σκυλακάκη, σύντομα παρακαλώ γιατί ξεπεράσαμε το χρόνο. Η ερώτησή μου, η συμπληρωματική μου ερώτηση είναι θα μπορούσατε να κάνετε το ίδιο χωρίς να είχατε κάνει αυτές τις δηλώσεις δημόσια σε μια συνέντευξη τύπου. Θα μπορούσατε να περιμένατε ήσυχα μέχρι να ξεκινήσει η δικαστική διαδικασία. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν να αντισταθεί κανείς στον τύπο. Είναι αδύνατον. Και δεν θα ήταν και σωστό και δίκαιο. Πώς θα βλέπατε εσείς έναν επίτροπο να παρετείτε εξαιτία μιας ε, διερεύνησης από μέρους Όλαφ ή δε Όλαφ να σιωπά. Μα για λόγους διαφάνειας δεν είμαστε σε μια μυστική υπηρεσία. Και σε αυτή την περίπτωση θα είχαμε κατηγορηθεί για έλλειψη διαφάνειας και εν δεν μπορούσα να πω τίποτα παραπάνω όσον αφορά το περιεχόμενο αυτής της ε, έκθεσης, αυτής της έρευνας, διότι υπήρχε η, ε, ο απαραίτητος σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας. Έπρεπε λοιπόν να κάνουμε κάποιες δηλώσεις, καθότι η σιωπή μας θα είχε ερμηνευθεί ως έλλειψη διαφάνειας και οι επιπτώσεις ήταν χειρότερες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Στάς, εκπρόσωπος των Πρασίνων, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Εκτός μικροφώνου. Eh, Η τεχνολογία, τι να κάνουμε. Κύριε Κέσλερ, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή τις απαντήσεις που έχετε μέχρι τώρα δώσει σε ερωτήσεις μας. Δεν μπορώ όμως να πω ότι είμαι απόλυτα ικανοποιημένος ε, μέχρι στιγμής. Νομίζω ότι υπήρξαν και κάποιες προσπάθειες από προσανατολισμού μας. Μας δόθηκαν λάθος πληροφορίες ενδεχομένω, όπως το 93C. Για την ε, κυρία Σεμπρί, ξέρετε ότι ήταν και μέλος ε, της Επιτροπής ε, της Έρευνας τέσσερις συνεντεύξεις που έχουν γίνει έγιναν ε, παρουσία της ε, στη Μάλτα τον ε, κύριο Ζάμι όταν τον ρωτούσαν εκεί αυτή τέλειωσε χρέη διερμηνέως άρα δεν μας έχουν πει την αλήθεια για όλα But I, I'm not sure I understand. I understood the, uh, the issue that we didn't say the truth. Anyway, I will tell you what has. Κοιτάξτε, θα σας πω εγώ τι συνέβη και εσείς μπορείτε να αποφασίσετε αν δεν είναι αλήθεια ή όχι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο. Η κυρία Σέμπρη, η Σκέμπρη, δεν ξέρω πώς προφέρεται, ήταν ε, διευθύντρια του γραφείου της Μάλτας, ε, που είναι το ομόλογο γραφείο για την καταπλέμψη ε, στη Μάλτα. Συνήθως συνεργαζόμαστε με τους εθνικούς φορείς ε, κατά πολέμης απάτης στη χώρα μας. Τι έγινε με τις ε, έρευνες που κάναμε στη Μάλτα. Μόνο για αυτές, μόνο για αυτές ήταν παρουσία της ε, κυρίας Έμπρη. Είπατε κάτι για συνεντεύξεις όταν τέσσερις, τέλος δεν το ξέρω αυτό. Τον κύριο Σίλβιο Ζάμι, τα πράγματι παρουσία της κυρίας Σέμπρη το κάναμε ερωτήσεις στη Μάλτα. Είχαμε συνεντεύξει οι οποίε έγιναν και στα ίδια τη γραφεία τη ΑΦΚΟ, τη ε, Μαλτέζικη Υπηρεσία δηλαδή, κατά πολέμου απάτη. Έτσι συνηθίζεται άλλωστε. Και εκεί είχαμε και μία συνέντευξη με τον κύριο Γκέιλ Κίμπερλι στην Μάλτα, στα γραφεία τη ΑΦΚΟ, παρουσία τη διευθύντρια ε, του οργανισμού. Δεν το παραδέχομαι λέγοντα ότι είναι κάτι κακό ή ότι είμαι ένοχο για κάτι είναι καταγεγραμμένο και στα πρακτικά των συνεντεύξεων, ήταν σαφές διότι έλαβε μέρος εκεί και έχει γραφεί και το όνομά της στα πρακτικά, τα έχει υπογράψει. Μιλώ για τις συνεντεύξεις ήταν παρούσα, δηλαδή τις συνεντεύξεις οι οποίες έλαβαν χώρα στη Μάλτα, στα γραφεία τη μαλτέσικη Υπηρεσία καταβολή Απάτη. Τώρα, κατά πόσον ε, ήταν διερμίαση, ή όχι. Τι να σα πω, σε κάποιε περιπτώσει έγιναν στα αγγλικά οι συνεντεύξει. Όλε οι συνεντεύξει έγιναν στα αγγλικά. Μια γλώσσα ευρέω διαδεδομένη που χρησιμοποιείται ευρέω και τη χρησιμοποιούν πολύ καλά και ο κύριος Ζάμιτ και ο κύριος Γκέμπριλ κυρία Σέμπρη, νομίζω, από ό,τι θυμάμαι τουλάχιστον, βοήθησε απλά στη μετάφραση κάποιων εκφράσεων από τα Μαλτέζικα στα Αγγλικά. Ένα λεπτό, μία δεύτερη ερώτηση από τον κύριο Στάση. Ευχαριστώ. Στην σελίδα 31 του ερωτηματολογίου, στις απαντήσεις για την 93C, για την κυρία Σέμπρη, λέτε ότι δεν ήταν παρούσα στις συνεντεύξεις, αλλά στις ε, ανακρίσεις. Μήπως λέτε κάτι διαφορετικό εδώ, προσπαθείτε να μας παραπλανήσετε, τι γίνεται. Δεύτερη συμπληρωματική ερώτηση. Λέτε, she was not present at the interview, she played no role in the whole investigation. Λοιπόν, το δεύτερο, Πώς γίνεται ένας άνθρωπος τρεις φορές ταυτόχρονα να δέχεται συνέντευξη, δηλαδή με κλόνους ε, εργάζεστε, πώς γίνονται οι συνεντεύξεις να είναι ταυτόχρονες, τρεις. Ή μας ε, είναι μια συνωμοσία όλα αυτά για να μας ε, κοροϊδέψετε. Κύριε και ένα λεπτό έχει το λόγο. Επαναλαμβάνω ότι η κυρία Σέμπρη συμμετείχε σε τρεις ή δύο τέλος πάντων συνεντεύξεις που έγιναν στα γραφεία της Περισκαταπολέμησης Απάτης στη Μάλτα. Έχουν καταγραφεί και στα πρακτικά. Δεν συμμετείχε στην έρευνα όμως συνολικά και δεν είχε κανέναν ρόλο για την κατάρτιση έκθεση ή για οτιδήποτε σχετικό. Απλά παρίστατο σε αυτές τις ε, συνεντεύξεις στη Μάλτα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερο. βλέπω να εκπλήσεστε κατά κάποιο τρόπο που κάποιοι πήγαιναν στις ε, σεντεκτό παραπάνω από ένα. Δεν είναι κάτι περίεργο. Θα σας αναφέρω όμως μια περίπτωση. Τι έγινε. Στις πρώτες συνεντεύξεις που κάνουν στο πλαίσιο της έρευνας, οι πρώτες ήταν συνέντευξη από τη Swedish Match. Τώρα πόσοι ήταν δεν θυμάμαι, τρεις, τέσσερις. Τους καλέσαμε και ήρθαν στην Όλαφ, στα κτίρια της Όλαφ. Ταυτόχρονα. Γιατί το κάναμε ταυτόχρονα, για να εγγυηθούμε την γνησιότητα, την αυθεντία των απαντήσεων, των συνεντεύξεων. Και για να αποφύγουμε, επειδή αν ε, έχουμε ουσιαστικά ε, τις ερωτήσεις προς τον ένα, μετά προς τον δεύτερο, μετά προς τον τρίτο, μπορεί κάπως να υπάρξει μια ενημέρωση για τις ερωτήσεις, για το τι απαντήσεις μπορεί να δώσει επόμενος και τα λοιπά. Θέλαμε να το αποφύγουμε λοιπόν αυτό, να υπάρχει μια συμφωνία μεταξύ τους για το τι, αποφάσι, ε, τι απαντήσεις θα δώσουν ή να ενημερώνει ένας τον άλλο για τις ερωτήσεις που τετέσει και τις απαντήσεις που έδωσε. Γι' αυτό και έγινε ταυτόχρονα η συνέντευξη το καθενός, ε, δηλαδή στο ίδιο όροφο σε τρία-τέσσερα διαφορετικά γραφεία. Διαφορετικοί ήταν ε, οι ανακριτές σε κάθε περίπτωση. Ο ένας που είναι και ο επικεφαλής Τώρα πάντα και δύο δεν ξέρω. Πάντως ένα σίγουρα. Ε, αυτό μπορώ να σα πω τι έκανε. Συμμετείχε σε πάνω από μία συνεντεύξη, ο ένας αυτό που θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, γιατί έπρεπε να εξασφαλιστεί ότι οι ερωτήσεις που θα υποβάλαμε στους ε, συνδευξεζόμενους από τη ειδικοί μάτς θα μπορούσε να ενημερώσει αυτός ε, τους ε, ανθρώπους μας που έκανε συνεντεύξεις στις, στα άλλα γραφεία για να τους κάνουν αντίστοιχες ερωτήσεις και να τους ενημερώσει και για τις απαντήσεις. Δεν ε, είναι τίποτα περίεργο, ούτε κανένα θαύμα. Πήγαινε αυτός ο ανακτής από το ένα γραφείο στο άλλο για να φροντίσει να τεθούν οι σωστές ερωτήσεις από όλους τους ερωτώντες. Η συμμετοχή του αν σε κάθε συνέντευξη και βέβαια επειδή μα θέλαμε να είμαστε απόλυτα σωστοί, κατεγράφει η παρουσία του σε αυτέ τις συνέντευξει. Δεν έγινε τίποτα κρυφό. Κυρία Αντρέας, τώρα έχει το λόγο από την ομάδα ECR. Για ένα λεπτό. Thank you, Chair. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επαναλάβω ότι δεν είμαστε εμείς ε, ερευνητική επιτροπή και δεν μπορούμε να μπούμε στις λεπτομέρειες της ερευνητικής διαδικασίας γιατί δεν καλύπτεται αυτό από την εντολή μας. Όμως έχω κάποια μελήματα, ανησυχίες όσον αφορά ε, την ε, ε, ανεξαρτησία της Όλαφ, ανησυχίες που διαρκούν 10 χρόνια η Όλαφ μπορεί να ξεκινήσει ε, διερεύνηση εάν υπάρχει εσωτερική, εσωτερικό πρόβλημα ε, με κάποιον υπάλληλο ή εργαζόμενο. Ε, άρα είναι νόμιμη η ανάμειξη της Όλαφ. Πόσες φορές όμως στέλνει η Όλαφ περιπτώσεις προβλήματος με θεσμικά όργανα. Επίσης, Γνωρίζετε ότι εάν, ε, γνωρίζετε αν ο, ο Επίτροπος Ντάλι έχει ε, υποβάλει ε, οποιαδήποτε διαδικασία προσφυγής και έχουν καταπατηθεί τα δικαιώματά του όσον αφορά αυτό το δικαίωμα που έχει ο κύριος Κέσλερ. Δεν ξέρω αν σας κατάλαβα καλά. Τι ρωτάτε, εάν η Κομισιόν μας έχει στείλει και άλλες πληροφορίες ή, κάποιες, ή, ή άλλες προσφυγές η Κομισιόν είναι ένα μεγάλο ε, σώμα. Από τους γενικούς διευθυντές της Κομισιόν, ναι βεβαίως, πολλές προσφυγές και αιτήματα και μάλιστα υποχρεούνται, υποχρεούνται δια του κανονισμού ε, να ζητήσουν διευκρινήσεις ε, και η διερεύνηση από την Όλαφ για περιπτώσεις ε, είτε υποψίας απάτης είτε σοβαρών ε, ατοπιμάτων συμπεριφοράς ε, ε, υπαλλήλων. Αυτό που διεφάνει σαφώς και φαίνεται άλλωστε και από την τελευταία ετήσια έκθεση της Όλαφ είναι ότι από πέρσι, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, από πέρσι έχουμε δει μία αυξητική τάση αυτών των υπονοιών. που στέλνουν στην Όλαφ όχι μόνο η Κομισιόν αλλά και τα άλλα ενωσιακά θεσμικά όργανα. Έχουμε ε, σταθερή αυξητική πορεία στα τελευταία χρόνια. Και από πέρσι μέχρι φέτος πάλι είδαμε μεγάλη αύξηση των ε, περιπτώσεων αυτών. Ζητείτε λοιπόν από την Όλαφ ε, διαφάνεια και στην αντιμετώπιση αυτών των ε, υποθέσεων. Και η δεύτερη ερώτησή σας, μπορείτε να μου τη θυμίσετε ποιο ήταν το δεύτερο σκέλος. Α, εάν έχει κάνει προσφυγή ο κύριος Ντάλι ή αν έχει υποβάλει παράπονα. Κοιτάξτε, ε, κάθε φορά που ήθελε να εκφράσει κάποια ανησυχία ή κάποιο παράπονο ε, ε, το έκανε μέσω του τύπου. Αλλά πρέπει να σας πω ότι έχει υποβάλει προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου κατά της Κομισιόν κατά της ε, Κομισιόν για μία σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τούτη την υπόθεση Και όσον αφορά την Όλαφ, επίσης έχει αναφέρει το γεγονός ότι παρακάμψαμε την Επιτροπή Εποπτείας στην διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό είναι, ε, ε, ε γι' αυτό κατηγορεί την Όλαφ, τουλάχιστον αυτό έχει υποπέσει στη δική μου ε, αντίληψη. Ε, ζητώντας και από τον τότε πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας κύριο Τίμενμανς ε, να ε, είναι μάρτυρας για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε συμπληρωματική ερώτηση. Θα ήθελα να διευκρινίσω αυτό που άκουσα. Στην <clears throat> αυξητική αυτή τάση που λέτε όσον αφορά τις προσφυγές. Αυτό συνέβη από την υπόθεση Ντάλι και μετά ή είχε παρατηρηθεί και πριν την υπόθεση Ντάλι αυτή η αύξηση των προσφυγών. Δεύτερον, τι σας προσάπτει ο Επίτροπος Ντάλι ότι παρακάμψατε την Επιτροπή Εποπτείας ή ότι παραβιάσετε τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Κοιτάξτε, όταν αναφέρθηκα σε αυτή την αύξηση των περιπτώσεων που έχουν λάβει και η Επιτροπή, αναφερόμουν σε όλο το έτος 2012, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχω συγκεκριμένες στατιστικές για αύξηση πριν ή μετά την υπόθεση Ντάλι, πριν δηλαδή τον Οκτώβριο ή μετά τον Οκτώβριο του 2012 δεν μπορώ να σας δώσω μια τόσο συγκεκριμένη αν θέλετε απάντηση. Τώρα, το δεύτερο ερώτημα. Από ό,τι ξέρω, ίσως να έκανα και κάτι που δεν το γνωρίζω, αλλά από ό,τι ξέρω παραπονέθηκε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά του παραβιάστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της έρευνας, γιατί παραβιάσαμε την Επιτροπή Εποπτείας και στείλαμε κατευθείαν την υπόθεση στις βελγικές αρχές. Ευχαριστώ πολύ. Ο εκπρόσωπος της Γκούε είναι ο κύριος Ντεγιούγκ σήμερα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Όταν εξετάσει κανείς το σύνολο της υπόθεσης Ντάλι, έχει την εντύπωση ότι υπήρχε μια πίεση για επιτάχυνση της διαδικασίας και αυτό οδήγησε σε μια μεγάλη σειρά σφαλμάτων ε, από μέρους της Όλαφ. Το θέμα τώρα είναι, κύριε Κέσλερ, ποιες εγγύσεις υπάρχουν στην υπηρεσία σας, όχι μόνο για σας, για τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της Όλαφ. Και μπορεί κανείς να αγνοήσει κάποιες από τις ε, αιτήσει της Επιτροπής για να διασφαλιστεί αυτή η ανεξαρτησία. Κοιτάξτε, εμείς δεν είχαμε καμία οδηγία ή προσπάθεια επιρροής από κανέναν εξωτερικό φορέα, όπως ακούγεται πολλές φορές και διαβάζουμε στον τύπο. Είναι πολύ δύσκολο να υπερασπιστώ τον εαυτό μου αν δεν ξέρω τις κατηγορίες. Εγώ διάβασα πάντως επανειλημμένος και με δύο τρόπο ότι χρηματοδοτούμαστε από την κάπνο καπνοβιομηχανία. Αλλά αυτό είναι λάθος. Είναι αβάσιμο και εντελώς λανθασμένο. Και δεν υπάρχει απολύτως καμία απόδειξη για κάτι τέτοιο, για αυτή την κατηγορία. Τώρα όσον αφορά την Επιτροπή, καμία οδηγία δεν μας δόθηκε και απολύτως καμία πίεση δεν ασκήθηκε σε μας. Έχουμε ένα γράμμα, μια επιστολή της Κάτριν Day, μια επιστολή γνωστή και σε πλήρη διαφάνεια έγινε αυτό. Την επιστολή αυτή γράφει ότι φυσικά αυτό είναι θέμα προτεραιότητας. Εμείς δεν το θεωρούμε αυτό σαν περιορισμό της ανεξαρτησίας μας, αλλά το θεωρήσαμε σαν μία σύσταση που πραγματικά ακολουθεί την κοινή λογική τι να σας πω, πριν από δύο εβδομάδες λάβαμε και μια άλλη αίτηση για διερεύνηση μιας άλλης υπόθεσης και η επιστολή που μας εστάλει περιείχε τη φράση «Σας παρακαλώ πολύ να διεκπαιρεώσετε αυτή την υπόθεση μέσα σε 15 μέρες». Κάνουμε ό,τι μπορούμε και σε καμία περίπτωση τέτοιου είδους ε, συστάσεις δεν μας ε, φαίνονται σαν περιορισμός της ανεξαρτησίας μας. Αυτό που μας είπε η Επιτροπή είναι, είναι ένα σημαντικό θέμα και θεωρήστε το θέμα προτεραιότητας για την προστασία της φήμης της Επιτροπής. Αυτό σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει ότι βιαστήκαμε. Πέντε μήνες κράτησε αυτή η έρευνα θα μπορούσαμε να είχαμε διεκπαιρεώσει και πιο γρήγορα ακόμα αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα κάποιοι βουλευτές, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, μας κατηγόρησαν ότι αργούμε πάρα πολύ για τη διαδικασία που τους αφορούσε κράτησε πέντε μήνες. Δεν ακούμε την παρέμβαση. Κύριε Τιγιόγκ, μπορείτε να κάνετε μια συμπληρωματική ερώτηση για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, διαπιστώνω ότι δεν απαντήθηκε η πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ποιες είναι οι διασφαλίσεις ε, όσον αφορά τις διεργασίες και τις διαδικασίες στην Όλαφ. Δεν μου εδόθη απάντηση. Η δεύτερη ερώτηση, πώς διασφαλίζετε την ανεξαρτησία σας απέναντι στην Κομισιόν και επίσης ε, γιατί δεν διαμαρτύρεστε. Ε, εάν μου έδιναν σε μια τέτοια περίπτωση ε, μια επιστολή λέγοντας κατά προτεραιότητα να ασχοληθείτε με το θέμα αυτό, θα διαμαρτυρόμουν, θα έλεγα να κοιτάξετε τη δουλειά σας. Απάντηση. Κοιτάξτε, εγώ ούτε προσευλήθην, από τον ε, πρόεδρο Μπαρόζο που μου ζήτησε κατά προτεραιότητα να ασχοληθώ με το θέμα αυτό, ούτε και ενοχλούμε όταν ε, κάποιες άλλες, ε, κάποια άλλα θεσμικά όργανα μου ζητούν γρήγορα να αντιμετωπίσω κάποια ζητήματα που σχετίζονται με το προσωπικό τους, γιατί πρέπει και εκείνοι να πάρουν τα μέτρα τους. Όσον αφορά τώρα τις διασφαλίσεις, αυτές περιέχονται στον κανονισμό. Έχουμε ε, δικές μας ανεξάρτητες διερευνητικές ε, διαδικασίες, ε, οι οποίες περιλαμβάνονται στον κανονισμό της Όλαφ. Υπάρχει ένα άρθρο, το οποίο λησμονώ αυτή τη στιγμή, πάντως το παραθέτω στα γραπτά μου, στις γραπτές μου σημειώσεις. Ένα άρθρο λοιπόν που λέει ρητά ότι ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ μπορεί να ε, φτάσει στα δικαστήρια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν θεωρήσει ότι κλπ. κλπ. Ε, και άλλωστε η Επιτροπή Εποπτείας σε κύριο ρόλο έχει την προστασία της ανεξαρτησία της Όλαφ αλλά βεβαίως και τον έλεγχο της ιδίας αυτής ανεξαρτησίας μελέτησαν προσεκτικά την περίπτωση αυτή και δεν διεπίστωσαν κανένα, ε, καμία ένδειξη ε, έλλειψης ε, ανεξαρτησίας ή καταπάτησης ανεξαρτησίας Όλαφ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ιρεν Χάουζερ δεν είναι στην αίθουσα. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο δεύτερο γύρο των ερωτήσεων. Ποιος θα πάρει το λόγο για το ΕΛΚ πάλι, κυρία Κρέσλερ. Κύριε έχω μία ερώτηση κι εγώ. Είπατε, είπατε δύο φορές, επαναλάβατε δύο φορές, ότι είναι σαφές για σας ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σε αυτήν την έρευνα. Θεωρείτε ότι σας έχει καταλάβει σωστά ή όχι ο πρόεδρος Μπαρόζο. Θεωρείτε ότι έφτασε σε σωστά συμπεράσματα ο πρόεδρος Μπαρόζο ή όχι. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα δεν κρίνω αποφάσεις που έχουν λάβει άλλοι ή ε, οι πολιτικές αρχές. Δεν είναι ο ρόλος μου αυτός και δεν θα το κάνω. Δεν είμαι σε θέση και δεν πρόκειται να αξιολογήσω συμπεράσματα τα οποία έχουν ε, εξάγει πολιτικοί παράγοντες επί του προκειμένου. Αυτό που είπα σήμερα και αυτό που είπα και στην ε, συνέντευξη τύπου μετά την παρέτηση του Επιτρόπου. Είναι αυτό που, γράφει, που ε, είχε γραφεί και στην ε, έκθεση, δηλαδή ότι δεν έχουν υπάρξει αποδεικτικά στοιχεία αποδεικτικά στοιχεία τα οποία να αποδεικνύουν ότι ο κύριος Νταλή ε, ήταν ο ηθήνων νους ε, ή με κάποιο τρόπο διευκόλυνε ε, την διαδικασία την παράνομη In our understanding. την, την οποία έπραξε άλλος, ένα τρίτο άτομο. Αυτό γράφει στην ε, έκθεσή μας. No conclusive evidence, ε, δηλαδή δεν έχουν προκύψει ε, τελειωτικά αποδεικτικά στοιχεία για οποιαδήποτε ποινική ευθύνη του κυρίου Νταλή. Όλα τα υπόλοιπα θα κριθούν στη Μάλτα από την ποινική δικαιοσύνη. Όσον αφορά τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν σε πολιτικό επίπεδο ή τα συμπεράσματα τα οποία ε, ε, έγιναν σε πολιτικό επίπεδο δεν βασίστηκαν στο κατά πόσον υπήρξαν συγκεκριμένα αποδεικτικά στοιχεία για την ποινική ευθύνη του Υπουργού. Ελήφθησαν επί τη βάση πολιτικών θεωρήσεων. Μία αποσαφήνιση πολύ σύντομη. Η έκθεση της Όλαφ χρησιμοποιήθηκε στην πολιτική συζήτηση που σχετίστηκε και με την ε, αποχώρηση, αποπομπή μάλλον του κυρίου ε, Νταλή. Δεν θεωρείτε ότι από τη δική σας πλευρά θα έπρεπε να έχει καταστεί πολύ πιο σαφές ότι αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία στα οποία καταλήξατε δεν θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε οποιαδήποτε πολιτική συζήτηση. Απάντηση. Να σας πω λοιπόν ότι και στο γραπτό μου υπόμνημα αναφέρομαι διεξοδικότερα στο θέμα αυτό. Να πω πάντως το εξής. Οι πολιτικές αποφάσεις ελήφθησαν, τα πολιτικά συμπεράσματα εξήχθησαν από τους πολιτικούς πρωταγωνιστές ε, σε σχέση και βασιζόμενα με αδιαμφισβήτητα αποδεικτικά στοιχεία. Όχι ε, με βάση στοιχεία τα οποία αφορούν την δικαιοσύνη και θα κριθούν ενώπιον των δικαστηρίων. Η έκθεση της Όλαφ επέστησε την προσοχή όλων των εμπλεκομένων ε, σε διάφορα στοιχεία τα οποία ήταν σαφή, τα οποία προέκυψαν κατά διάρκεια της διερευνητικής διαδικασίας και αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν την Κομισιόν σε πολιτικές αποφάσεις όσον αφορά ε, το ζήτημα το οποίο σχετίζεται με τις πολιτικές ευθύνες του εν λόγω ατόμου και όχι με τις ποινικέ του ευθύνες. Τώρα η κυρία Γκρέσλε εκ μέρους της ΕΛΚ. Αυτό που είναι πολύ ιδιαίτερο με τη συζήτηση που έχουμε με τον κύριο Κέσλερ είναι ότι υπάρχουν μισές αλήθειες, περίπου αλήθειες και διάφοροι χειρισμοί της αλήθειας θα έλεγα. Αναφερόμαστε στις, ε, στα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία, έτσι όπως τα παρουσιάζει ο κύριος Κέσλερ με τον ορισμό circumstantial evidence, ε, δεν είναι ικανοποιητική. Είτε είναι αποδεικτικά στοιχεία είτε δεν είναι αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό που επίσης ε, με προβληματίζει σε σχέση με τις συστάσεις, πότε επιτέλους θα προετοιμαστούν με τρόπο έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να τις λάβουμε. Το ερώτημα επίσης που με προβληματίζει είναι γιατί δεν απαντήσατε στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 50% των ερωτήσεων δεν απαντήσαν. Αυτό είναι σκανδαλώδες. Και ουσιαστικά το ίδιο κάνετε και εδώ. Μισές απαντήσεις, μισές αλήθειες. Και αυτό που διαπιστώνω είναι ότι όταν υπάρχει πίεση, ουσιαστικά δεν μας απαντάτε και Αν θέλετε, στην ερώτηση για το φαγητό, για το γεύμα το οποίο, ε, για το οποίο σας κάναμε την ερώτηση είναι ότι και αυτό αποτελεί τμήμα της ερευνητικής διαδικασίας και αποτελεί τμήμα των στοιχείων. Για να δούμε λίγο τις ερωτήσεις με τη σειρά. That was ε, question number 36. Είναι η ερώτηση παριθμών 36 ή 37. 36B. Ναι. Τη βρήκατε? Άψογα. Αναφερθήκατε σε αυτά τα circumstantial evidence. Υπάρχουν αυτά και υπάρχουν και τα άμεσα στοιχεία. Δεν το εφήβρα εγώ αυτό το σύστημα. Όπως σαφώς και ρητά αναφέρεται στην έκθεση που σας έδωσα την αναφορά που σας έδωσα το πρωί, υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δεν σχετίζονται με την ποινική ευθύνη, αλλά κάποια άλλα ζητήματα τα οποία αποτέλεσαν βάση ε, για τα πολιτικά συμπεράσματα τα οποία εξήγαγαν ε, οι ε, πολιτικοί πρωταγωνιστές. Αυτά ήταν κάποια στοιχεία τα οποία σαφώς κατεδείχθησαν ε, και τα οποία, και τα οποία αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν είναι καν ε, αποδεικτικά στοιχεία, είναι στοιχεία, είναι δεδομένα επί των οποίων βασίστηκαν κάποια πολιτικά συμπεράσματα. Η κυρία Γκρέσλερ στη δήλωσή της έκανε αναφορά σε συστάσεις, εάν κατάλαβα καλά. Τις συστάσεις που έκανε η Όλαφ μπορώ να φανταστώ. Να σας πω λοιπόν ότι η Όλαφ δεν έκανε καμία σύσταση. Η Όλαφ έστειλε την ε, έκθεση στην Κομισιόν μαζί με μία ε, επιστολή όπου ρητά αναφέρεται και παραθέτω καταθέτουμε ε, το ζήτημα ε, σε εσά έτσι ώστε να το μελετήσετε και να λάβετε τις αποφάσεις σας ε, για τη συμπεριφορά του Επιτρόπου. Αυτή είναι η σύστασή μου αν μπορούμε να την ονομάσουμε έτσι δηλαδή για έλεγχο, για έλεγχο μιας ηθικά επιλήψιμης ή όχι και πολιτικά επιλήψιμης ή όχι συμπεριφοράς. Όσον αφορά το δικαστικό ζήτημα, να σας πω ότι εμείς δεν κάναμε καμία δικαστική φύσεως ε, πρόταση. Είπαμε απλώς ότι στέλνουμε τον σχετικό φάκελο στον Γενικό Εισαγγελέα της Μάλτας. Δεν ζητήσαμε την απαγγελία ε, κατηγοριών για οποιονδήποτε εμείς απλώς είπαμε υποβάλλουμε τον φάκελο ε, προς εξέταση από πλευρά σας και ενδεχόμενη δικαστική συνέχεια. Και επίσης κανένα στοιχείο δεν αποκάλυψα στον τύπο το οποίο δεν είχα αποκαλύψει σε εσά. Απαντήσαμε στις ερωτήσεις που, του ερωτηματολόγιου που μας στείλατε και επίσης ε, απήντησα και σε κοινοβουλευτικό ερώτημα ε, το οποίο είχατε υποβάλει με το ίδιο θέμα. Πάντα πρώτα σε εσά απαντούσαμε. Η κυρία Γκρέσλερ. Κοιτάξτε, στις 5 ε, Μαΐου αναφερθήκατε σε αυτό το γεύμα. Στις 5 Μαΐου απαντήσατε και κάποιες άλλες ερωτήσεις όσον αφορά το θέμα της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε και εδώ αναφέρομαι και στην ερώτηση 36π. Εδώ βλέπω όμως η απάντησή σας να είναι τελείως διαφορετική όσον αφορά την μαρτυρία αυτή. Κοιτάξτε, δεν έδωσα καμία συνέντευξη, καμία για το θέμα αυτό. την εφημερίδα Times of Malta. Τι είπα στη Malta Today, δεν ξέρω. Για το θέμα αυτό, στο Times of Malta, α, είπα τα ίδια. Τα ίδια ακριβώς που, που είχα πει απαντώντας ε, στην ερώτηση του βουλευτού επιτρέψτε μου σαν πρόεδρος να διαπιστώσω ότι δεν απαντήθηκε το ερώτημα ούτε για τα έξοδα τα ταξιδιωτικά, ούτε για το γεύμα. Κοιτάξτε. Για θέμα τέτοιο δεν μίλησα σίγουρα ε, εξόδα μετακίνηση, εξόδων ταξιδίου για τα έξοδα αποστολή ε, στις ε, έρευνες αυτές. Ε, είναι σαφή τα πράγματα. Εμείς το συζητήσαμε και με τους δικηγόρους μας όταν χρειάστηκε να απαντήσουμε τα περί εξόδων αποστολής στο ερωτηματολόγιο. Εγώ ήμουν υπέρ του να απαντήσω γιατί το να μην απαντήσω θα ήταν σαν να είχα κάτι να κρύψω. Αλλά βέβαια πολύ σωστά οι δικηγόροι μας επισήμαναν το εξή. Εάν αρχίζουμε να αποκαλύπτουμε πράγματα, πλέον όχι στο κοινοβούλιο, αλλά στον τύπο και παντού, σε μια, στο πλαίσιο μια έρευνα η οποία είναι ακόμη σε εξέλιξη, γιατί αυτό είναι το, έτσι είναι τα πράγματα. Στη Μάλτα συνεχίζεται η δραστηριότητα αυτή της έρευνας. Οπότε θα ήταν σαν μέχρι εκ των προτέρων αποκάλυψη των ερευνών και των αποτελεσμάτων και αυτό σίγουρα ε, ή θα μπορούσε τέλο πάντων να παρακολύσει την συνεχιζόμενη έρευνα ενώπιον των δικαστηρίων. Δεν υπάρχει τίποτα περίεργο. Αν δείτε με τις συνεντεύξεις πρώτα καταλάβετε που έγιναν οι αποστολές, που έγιναν οι συνεντεύξεις. Φαίνεται από τον τόπο της διεξαγωγής της συνέντευξης. Αλλά είναι θέμα αρχή, γιατί θέτουμε προηγούμενο. αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Δηλαδή, το προηγούμενο τότε αποκαλύπτονται δημοσία όλες οι πράξεις ε, έρευνας ε, που διεξάγουμε, γιατί αυτό μπορεί να βλάψει, να παρακολύσει την όλη έρευνα, αν εκ των προτέρων αποκαλύψουμε τις δραστηριότητε αυτές. Κοιτάξτε, δεν βλέπετε αντίφαση. Απαντήσατε στο Times of Malta, στην εφημερίδα αυτή, και δεν απαντάτε εδώ, στο Κοινοβούλιο. Συναντηθήκατε, ναι ή όχι, και διπνήσατε με τον μάρτυρα. Κοιτάξτε, δεν απάντησα στο Κοινοβούλιο όσον αφορά τα έξοδα του, της μετακίνησης. Ρωτήθηκα και δεν απάντησα. Ούτε στον τύπο, ούτε στο Κοινοβούλιο. Το θέμα του γεύματος ή του δείπνου απάντησα. Διότι η Όλαφ έτσι κι αλλιώς έκανε μια δημόσια δήλωση μετά από την διαρροή που έγινε από την Μάλτα. Αυτό είναι κάτι που προέκυψε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενώπιον των δικαστηρίων στην Μάλτα. Μετά από, επαναλαμβάνω, διαρροές και μετά από κάποιες πολύ μερικές διαρροές πληροφορίες. Πρόκειται λοιπόν για κάποιον για κάποιον που έκανε αυτές τις δηλώσεις μετά από την συνέντευξη που μας έδωσε. Και ουσιαστικά υπάρχουν ε, οι δηλώσεις στον τύπο που ε, αποσαφηνίζουν αυτό, γιατί νιώσαμε ότι έπρεπε να το κάνουμε. Και βεβαίως κατά τη διάρκεια της ε, συνέντευξης αυτής η μάρτυρας ήταν δυόμιση το απόγευμα όταν τελείωσε η συνέντευξή της. Προετοιμάζαμε, αν θέλετε, τα πρακτικά και ουσιαστικά τη ρώτησα αν ήθελε να ε, φάει κάτι. Την συνόδευσα λοιπόν, επρόκειτο για ένα διάλειμμα μισής ώρας. Τι να σας πω, δεν ήταν καν ε, γεύμα. Ήταν δυόμιση το μεσημέρι. Ήμασταν, αν θέλετε, για μισή ώρα κάναμε μια διακοπή για να φάμε κάτι. Γύρισε μετά, έκανε κάποιες αλλαγές, υπέγραψε και κατόπιν άλλες δύο φορές παρουσία δικηγόρου κατέθεσε σαν μάρτυρας. Και πρέπει να σας πω ότι αυτή είναι η ιστορία, αυτές ήταν οι διαρροές από μέρους της Μάλτας και εμείς σε, μια, σε ένα ανακοινοθέν τύπου ξεκαθαρίσαμε αλλά και σαν απάντηση σε μία από τις ερωτήσεις που μας έθεσε το Κοινοβούλιο και δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία αντίφαση. Πάρα πολύ σημαντικό λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποσαφήνισή σας. Μα δεν ήταν θέμα διαρροής. Τα είπε στο δικαστήριο αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαλτίζης. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά την ε, διεξαγωγή της συνεδρίασής μας, ε, πρέπει να πω ότι δεν αισθάνομαι ε, άνετα έχουμε ο καθένας δικαίωμα να θέσουμε δύο ερωτήσεις. Εδώ πρόκειται για τη δουλειά μας. Περίπτωση του κυρίου Νταλή πλέον αποτελεί υπόθεση στο δικαστήριο, οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Και αυτό το οποίο εμείς κάνουμε εδώ θα μπορούσε να θεωρηθεί ως παρέμβαση στο έργο της δικαιοσύνης. Δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε εμείς όμως ε, τα δικαστήρια. Ένα αυτό. Δεύτερον, το ζήτημα είναι άκρος πολύπλοκο. Είναι αυτονόητο αυτό. Δεν είναι μυστικό ότι ο γενικός διευθυντής ή οι άλλοι υπεύθυνοι ε, μπορεί να πάνε και σε άλλους φορείς να πούνε ακριβώς τα ίδια. Η Επιτροπή μας στο μέλλον Νομίζω ότι θα πρέπει να ασχοληθεί περισσότερο με την αποτελεσματική αξιοποίηση των χρημάτων των φορολογουμένων και ίσως να μην παρεμβαίνουμε τόσο σε αυτές τις γενικές συζητήσεις με βάση κάποια πολιτικά κίνητρα. Τέλος πάντων, το ερώτημά μου είναι το εξής. Η Όλαφ είναι ανεξάρτητος φορέας που διεξάγει έρευνες δικαστικής φύσεως θα έλεγα. Δεν ξέρω αν ε, θα μπορούσατε ενδεχομένως και με τους επιτρόπους, ε, τον Επιτρόπο των Αρμόδιων να συζητάτε κάποια θέματα για να μην δημοσιοποιούνται. Το θέμα είναι να υπάρχει ένα σύστημα για να αποφύγουμε υποθέσαν αυτή που μας απασχολεί εδώ και μήνες. Για δύο λεπτά First Πρώτα απ' όλα για τις πρώτες σας παρατηρήσεις κύριε Μπαλτσίτης. Με τις αρχές σας παρατηρήσεις συμφωνώ απόλυτα. Ως προς το ερώτημα, το τελευταίο. Το ερώτημα της κυρίας Γκρέσλι. Πολύ σωστά είπε ότι αυτά τα οποία είπε η Γκέιλ Κίμπριλ τα είπε στο δικαστήριο. Υπερασπιζόμουν τον εαυτό της τα είπε. Δεν βλέπετε να υπάρχει εδώ μια έλλειψη ισορροπίας, δεν βλέπετε κινδύνους, δεν βλέπετε ότι κινδυνεύουμε να θέσουμε ένα προηγούμενο. Εγώ δεσμεύομαι να απαντήσω σε αυτά τα οποία είπε και να τα αντικρούσω. Στα όσα είπε η ίδια στο πλαίσιο τη δίκη, τη διαδικασία, στο δικαστήριο. Και κατά κάποιο τρόπο τα είπε υπερασπιζόμενη ε, αυτήν. Και εγώ απαντώ εδώ. Δεν είναι περίεργο. Δεν υπάρχει προηγούμενο για κάτι τέτοιο και είναι και επικίνδυνο, ψοκίνδυνο ω διαδικασία. Νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε υπόψη. Προσεβασμό προς το Κοινοβούλιο απαντώ. Αλλά τελικά τι γίνεται, έχουμε δύο παράλληλες διαδικασίες. Κατά πάσα πιθανότητα για την ίδια ερώτηση ε, θα τεθεί το θέμα και στη Μάλτα, στο δικαστήριο. Ξέρει η ίδια τι γίνεται εδώ, τι λέμε εδώ, είμαι υπεύθυνο για αυτά που λέω εδώ. Παρακαλώ να έχετε υπόψη σας τις επιπτώσεις αυτού που κάνουμε. Είναι πολύ λεπτό το ζήτημα και ως ένα βαθμό η άσκηση αυτή, το εγχείρημα αυτό είναι και λίγο ρηψοκίνδυνο. Δηλαδή τι κάνουμε, απαντούμε σε διαρροές της ε, δίκης στη Μάλτα. Αυτά τώρα σε ό,τι αφορά το ερώτημα του κ. Μπαλτσίτης. Έχουμε ένα πλαίσιο για την πρακτική συνεργασία. Δεν ισχύει για μας, και για όλους τους οργανισμούς και το επικαιροποιούμε. Και με την Κομισιόν ε, έχουμε ρυθμίσει εργασίας για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών από δική σου πλευρά σε περίπτωση που έχουμε σοβαρές ε, αντιδοντολογικές συμπεριφορές, ε, τα κτλ. Και εμείς επίσης δίνουμε πληροφορίες και το ίδιο συμβαίνει και με άλλους οργανισμούς και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει ένα πλαίσιο για την καλή συνεργασία των θεσμικών οργάνων όταν έχουμε μια έρευνα σε εξέλιξη. Εξ όσο γνωρίζω, εντός Κομισιών, βέβαια είναι εκτός δικής μου, δικού μου πεδίου αρμοδιοτήτων, νομίζω ότι υπάρχει ε, κώδικα συμπεριφοράς, κώδικας διοντολογίας για την Κομισιόν, για τους επιτρόπους. Έχουμε κάνει και τη σχετική παραπομπή. Πριν από δύο χρόνια η Κομισιόν ε, έχει εγκρίνει και την ε, στρατηγική καταπολέμηση της απάτης που συμμετείχαμε και εμείς. Όπως και όλες οι γενικές διευθύνσεις της Κομισιόν. Είναι πολύ καλό αυτό το σύστημα και ίσως γι' αυτό και τον τελευταίο χρόνο ο αριθμός υποθέσεων ε, που φτάνουν στην θα έχει αυξηθεί. Ευχαριστώ. Κύριε Μπαλτσίτη, συμπληρωματική ερώτηση. Ένα λεπτό έχετε. Η ερώτησή μου ήταν απλή, πολύ απλή. Και η συμπληρωματική επίσης θα είναι απλή. Έχετε κοινή ε, στρατηγική με τον αρμόδιο ευρωπαϊκό Επίτροπο έτσι ώστε να αποφύγετε τέτοιου είδους ευαίσθητα ζητήματα να μην μπορούν να στραφούν ή να χρησιμοποιηθούν εναντίον τη ΟΛΑΦ. Γιατί ακούσαμε και σήμερα ότι έχουν υπάρξει διαρροές πληροφοριών και ε, αυτές οι διαρροές δεν θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά της ΟΛΑΦ ως ε, υπηρεσία ή θεσμού Ευχαριστώ κύριο Σκέφλερ, ένα λεπτό. Όχι, δεν υπάρχει ειδική στρατηγική από αυτού. Και ε, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αρμόδιο επίτροπο γιατί ο επίτροπος μας, ο, ο κύριος Σεμίτα, δεν είναι ε, υπεύθυνος για οποιασδήποτε διαρευνητικές διαδικασίες, ούτε αναφερόμαστε σε αυτόν την προκείμενη περίπτωση. Ναι, είναι πολιτικός υπεύθυνο για τις δραστηριότητε της Όλαφ, οι οποίε οι όμως δεν ε, ε, είναι οι διαρευνητικέ διαδικασίες αυτού του είδου οι ε, ανακρίσει και οι διερευνητικέ διαδικασίες αυτές. Εμείς αναφερόμαστε στον αρμόδιο επίτροπό μας, κ. Σεμίτα, για τις εν γέννη διαδικασίες μας. Τώρα, επί του προκειμένου, μπορέσαμε να κάνουμε μία πολύ λογική ε, και διεξοδική μελέτη, ε, έρευνα μάλλον, που διήρκεσε πέντε μήνες. Δεν και λίγο πέντε μήνες, χωρίς καμία διαρροή. Πήραμε βεβαίως όλα τα απαραίτητα μέτρα, τις απαραίτητες προφυλάξεις και επιτύχαμε να μην έχουμε καμία διαρροή που θα είχε ζημιώσει σοβαρότατα και τον εμπλεκόμενο επίτροπο και την επιτροπή στο σύνολό της. και ξέραμε ότι ο τύπος ήθελε πολύ να υπάρξουν διαρροές. Γι' αυτό προσέξαμε περισσότερο. Ένα λεπτό για την Άλντε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε απάντηση ερώτηση του κύριου Κάλβιν, ο κύριος Κέσσερ είπε ότι ε, εάν προέκυπτε παρόμοιο ζήτημα και αν είχαμε την επιλογή θα ξανακάναμε τα ίδια ακριβώς πράγματα. Παρατήρηση από αυτού. Ένα θέμα που με απασχολεί ακόμα είναι ότι η Όλαφε είναι Επιτροπή Επιτήρησης ε, και δεν ακολούθησε τις διαδικασίες που προβλέπεται από, τις, ε, από τον κανονισμό και νομίζω ότι αυτό το ανέφερε και ο κύριος Ντάλι ενώπιον του δικαστηρίου. Ο κύριος Κέσλερ θεωρεί ότι θα ήταν χρήσιμο εν τέλει να δώσει στην Επιτροπή Εποπτείας ε, την ευκαιρία να γνωμοδοτήσει ε, σε ιδιαίτερα ευαίσθητες περιπτώσεις ε, όπως ε, τούτη εδώ. Γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία πολιτικώς είναι ιδιαίτερο ευαίσθητα και επομένως μια ελάχιστη προφύλαξη θα ήταν να έχει τη δυνατότητα η Επιτροπή Εποπτείας να εκφραστεί. Δεύτερη ερώτηση. Η σχέση με την Επιτροπή Εποπτείας αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε ή όπως θα ήθελε. Ένα λεπτό κύριε Κέσλερ, ξανά να πούμε ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται ενώπιον του δικαστηρίου και χαίρομαι που είναι εκεί γιατί ε, ε, ε, εκεί θα ληφθεί η τελεσίδικη απόφαση την οποία θα πρέπει να σεβαστούμε όλοι με μένα πρωτον Αυτό που κάναμε με την Επιτροπή Εποπτείας σε αυτή την περίπτωση είναι απολύτως ευθυγραμμισμένο πρώτον με τον κανονισμό άρθρο 11 το οποίο ρητά αναφέρει ότι πρέπει να πληροφορήσουμε, inform στα αγγλικά, να πληροφορήσουμε την Επιτροπή Εποπτείας για τα ε, ε, ζητήματα, για τις υποθέσεις μάλλον οι οποίες ε, θα μεταφερθούν στα εθνικά δικαστικά συστήματα. Έχουμε μάλιστα το προηγούμενο της απόφασης του 2004, όπου το δικαστήριο ε, είπε να πληροφορείται η Επιτροπή Εποπτείας σημαίνει ότι θα πρέπει εκ των προτέρων να, τους, ε, να έχουν την πληροφόρηση πριν σταλεί το ζήτημα επομένως στη δικαστική διαδικασία. Η Όλαφ έχει καθιερώσει μια πρακτική η οποία είναι η εξής. Στέλνουμε τις υποθέσεις στην Επιτροπή Εποπτείας πέντε μέρες πριν τις στείλουμε στις εθνικές δικαστικές αρχές, εκτός και αν υπάρχουν ε, επίγουσες διαδικασίες. Πέντε ε, ημέρες πριν, που δεν είναι υποχρέωση που απορρέει από τις συνθήκες ή από τον κανονισμό, αλλά ε, ε, είναι μια πρακτική την οποία εμείς έχουμε καθορίσει. Μερικές φορές εάν υπάρχει κατεπίγουσα διαδικασία μπορεί αυτή η πενταήμερη, πενθήμερη συγγνώμη, ε, διορία να είναι μικρότερη. Και το Σεπτέμβριο λοιπόν εμείς γράψαμε σε γενικές γραμμές, στέλνουμε την πληροφόρηση της υπόθεσης πέντε μέρες πριν. Σε τούτη την περίπτωση στείλαμε την πληροφόρηση τρεις μέρες πριν, διότι το ζήτημα ήταν ήδη γνωστό ενώ σε άλλες περιπτώσεις ε, δεν γνωρίζει καθόλου το ζήτημα ε, ε, ο τύπος ή δεν έχει γνωστοποιηθεί το θέμα. Τη στιγμή όμως που ο Επίτροπος είχε παρετηθεί, το ζήτημα έγινε απολύτως γνωστό και επομένως εμείς επιλέξαμε τις τρεις μέρες και καλύπτεται αυτή η τριήμερη προθεσμία από τον κανονισμό που αναφέρει γενικά in advance, εκ των προτέρων, πριν σταλεί στις δικαστικές αρχές. Σεβαστήκαμε λοιπόν τον ε, κανονισμό. Μου είπατε επίσης ε, γιατί ε, δεν είχατε διαβούλευση. Πρέπει να ξέρετε ότι στην Επιτροπή Εποπτείας στέλνουμε 80 περίπου υποθέσεις τον χρόνο και η διαδικασία είναι πάντα ίδια. Τα στέλνουμε την πληροφόρηση, περιμένουμε πέντε μέρες, στην προκειμένη περίπτωση περιμέναμε, περιμέναμε ε, τρεις μέρες και μετά στείλαμε την πληροφόρηση στην δικαστική ε, αρχή σε αυτή την περίπτωση ενεργήσαμε όπως κάναμε και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις. Δεν θα μπορούσαμε σε τούτη την περίπτωση να τροποποιήσουμε τις διαδικασίες. Τις ακολουθήσαμε, τις σεβαστήκαμε και τις ακολουθήσαμε όπως σε κάθε άλλη περίπτωση. Ευχαριστώ. Ε, Συμπληρωματική ερώτηση στον κύριο Μούλτερ, δίνω το λόγο. Θα ήθελα να αναφερθώ στη σχέση που έχετε με την Επιτροπή Εποπτείας είναι ομαλή όπως την παρουσιάζει ο κύριος Κέσλερ. Εμείς όμως είχαμε άλλη εντύπωση μετά από την συνάντηση που είχαμε. Θα ήθελα να ξεκαθαριστεί το θέμα αυτό. Κύριε Κέσλερ, έχετε ένα λεπτό. Ναι, πράγματι, δεν απάντησα αυτό το ερώτημα. Κοιτάξτε, δεν είναι ιδεώδης. Ε, από δική μου πλευρά. βλέπω ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. και οι ίδιοι στην τελευταία συνάντηση εξέφρασαν ε, έλλειψη ικανοποίησης. Ε, αλλά είναι δύσκολη θέση μου κατά κάποιο τρόπο. Εγώ τηρώ αυστηρά τη συμφωνία που έχω μαζί τους. Δεν μπορούσα να κάνω άλλωστε και διαφορετικά, διότι πέρυσι το Σεπτέμβριο τα συμφωνήσαμε. Και μας είπαν ότι δεν τους ικανοποιεί αυτό. Τους είπα λοιπόν να μας πούν τι θέλουν να αλλάξει. Μας είπαν πριν δύο μήνες ήδη ότι θα γίνουν κάποιε αλλαγέ. Αλλά αν δεν μου πούνε εμένα ότι πρέπει να αλλάξω εγώ, δεν μπορώ να το κάνω από μόνο μου. Περιμένουμε λοιπόν. Συν ότι μετά την συνάντηση που είχαμε πριν από λίγες εβδομάδες ε, με την Επιτροπή Απτία στην Επιτροπή Κόντ, έδωσα έναν υπάλληλο παραπάνω, όπως είχαν αναγγείλει άρα έχουν το μέγιστο πλέον ε, προσωπικό που είχαν ε, μέσα στα τελευταία 14 χρόνια δεν έχουν αντιδράσει. Αυτό υποθέτω όμως ότι θα είναι ικανοποιημένοι. Δεύτερον, μετά τη συνάντηση, ο Επιτρόπος Σέμετα συγκάλεσε μία συνάντηση παρουσία αυτών και ε, μου για να δούμε ποια είναι τα θέματα επιτάπητος και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την ε, συνάντηση. Δεν δέχθηκε όμως η Επιτροπή Εποπτείας τη συνάντηση αυτή. Θα σας πει, είμαι βέβαιος, περισσότερο Επιτρόπος Έμετα. Ευχαριστώ. Ο εκπρόσωπος των Πρασίνων, ο κύριος Στάς, για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κέσλερ, θα ήθελα να επανέλθω στα ερωτήματα σε ό,τι αφορά ε, το γεύμα που είχατε με ένα μάρτυρα. λέγεται ότι η συνέντευξη κράτησε από τις 10 και ένα μέχρι τις 4.30 και λίγο παραπάνω. Και λέτε ότι ε, διακόψατε για γεύμα. Ε, πρώτον, κράτησε πολύ αυτή η που θέλετε. Και δεύτερο, φυσιολογικό να ξεκινάτε τη, ε, τη συνέντευξη, να διακόπτετε για δύο ώρες αφού φάτε κάτι και πιείτε κάτι με τη μάρτυρα. Είναι αυτό μια κανονική διαδικασία και θα, θα πρέπει να είναι πρακτικά. Και δεύτερον, Αν στόχος σας είναι με τις συνεντεύξεις να συγκεντρώσετε στοιχεία για να, όχι για, με στόχο την αθώση, αλλά την απαγγελή κατηγορία σε κάποιον τελικά. Και έχουμε και την αναθεώρηση της ε, οδηγίας για τον καπνό. Μπορούσαν να έχουν επιπτώσεις. Πάντως βλέπουμε ότι αθρώνονται οι ύποπτοι. Γιατί όλα αυτά τα τελευταία εξελίξεις για τη Μόζη Ντάλι δεν περιλαμβάνονται στη δική σας έκθεση. Κοιτάξτε, πολλές ερωτήσεις και έχω μόνο δύο λεπτά. Επανέρχομαι στο γεύμα. Όλες οι συνεντεύξεις με τους ε, μάρτυρες ε, από το Swedish Match, την Σίλβια Τάμιτ, όλους. Για όλους φάγαμε κάτι επιτόπου, μέσα στην αίθουσα. Κρουασάν, γλυκά, μπισκότα, αυτά είχαμε. Ήμασταν σε μία αίθουσα με την Γκέλ Κίμπερλι. Δεν είχαμε όμως τίποτα σε αυτή την περίπτωση. Είχε τελειώσει η συνέντευξη, ήταν δυόμιση. Δεν είχε όμως προετοιμαστεί το γραπτό κείμενο. Είχαμε περίπου 20 λεπτά, πεινούσε και μου είπε θα ήθελα να φάω κάτι. Και εγώ απλώς την συνόδευσα. Δεν επρόκειτο για μια δύο διακοπή, μισή ώρα. Κατόπιν γυρίσαμε, διάβασε την μαρτυρία της, η οποία ήταν πλέον έτοιμη, έκανε κάποιες αλλαγές και τελείωσε. Τίποτα παραπάνω. Είναι κάτι, αν θέλετε, που συμβαίνει, αν θέλει κάποιος να είναι ευγενής με αυτούς που είναι παρόντες, αν θέλει κάποιος να συμπεριφερθεί με ανθρώπινο τρόπο. Όχι. Δεν ήταν επιβαρυντική η συνέντευξη ήταν μόνο για να κατηγορήσουμε. Το γεγονός ότι διακόψαμε στο τέλος για μισή ώρα, μπορέσαμε να πάρουμε κάποιες πληροφορίες για μια συνάντηση με τον Επίτροπο. Και πριν ξεκινήσει η συνέντευξη, Νομίζαμε ότι αυτή η συνάντηση ήταν παρουσία της κυρίας Κίμπερλι. Κατόπιν διαπιστώσαμε ότι όχι, όχι και αυτό αναγράφεται στην έκθεση. Αντίθετα με αυτά που τελείως λανθασμένα αναφέρονται στον τύπο. <coughs> Αυτή η συνέντευξη λοιπόν κατά κάποιο τρόπο μείωσε αν θέλετε, αποδυνάμωσε τα στοιχεία, τα επιβαρυντικά στοιχεία, τα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά τις συναντήσεις του Επιτρόπου με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Συγκεντρώσαμε λοιπόν όλα τα στοιχεία υπέρ ή κατά. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν υπέρ, όπως αυτή που σας ανάφερα. Έχετε ένα λεπτό για μία επιπλέον ερώτηση. Διαπιστώνω ότι στις δυόμιση λέτε ότι διακόπη η συνάντηση. Εγώ διαβάζω όμως ότι αυτό έγινε στις δυόμιση. Πουθενά δεν λέτε ότι έγινε μια διακοπή. Και δεν απαντήσατε και στην ερώτησή μου, γιατί κάποια τμήματα αυτής της έρευνας δεν χρησιμοποιήθηκαν, ενώ ήταν ελαφρυντικά στοιχεία. Περίχανε ελαφρυντικά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη είναι η μαρτυρία του Διευθυντή της ε, Γενικής Διεύθυνσης ΣΑΝΚΟ που λέει ότι σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε επιρροή όσον αφορά την ε, τροποποίηση της οδηγίας για τον καπνό. Αυτό δεν το χρησιμοποιείται. Κάτι που τελικά έχει σαν αποτέλεσμα να καταρρεύσει η όλη σταδιοδρομία αυτού του Γενικού Διευθυντή. Το αναφέρεται στην έκθεση, είναι σαφές. Και παρεπιπτόντος, για τη σύντευξη τύπου που βλέπω τώρα ότι με ε, κατακρίνεται ότι έδωσα, πρέπει να σας πω ότι ακόμη και τη 17η του μήνα, δηλαδή μια-δυο μέρες μετά την παρέτηση του Επιτρόπου, συνέντευξη τύπου, βρήκαμε με την έρευνα της Όλαφ... ότι δεν έγινε καμία προσπάθεια, καμία απόπειρα αλλαγή τη νομοθεσία από τον Επίτροπο. Το είπα ξεκάθαρα σε αυτή τη συνέντευξη τότε και το λέει και η έκθεση. Δεν είναι δική μα έρευνα μόνο, δεν είναι μόνο η έκθεση. Υπάρχουν τα πρακτικά όλων των συνεντεύξεων, όλοι οι φάκελοι που έχουν όλοι σταλεί στι δικαστικέ αρχέ τη μάλτα. Όχι μόνο έκθεση. Στην Κομισιόν ΔΕ μαζί με την έκθεση επίσης αποστήλαμε όλες τις συνεντεύξεις. από τον Επίτροπο που ε, φυσικά υπερασπίστηκε αυτό. Όλα λοιπόν τα θεσμικά όργανα είχαν στη διάθεσή τους όλα τα στοιχεία. Είτε υπέρ του αν λόγω ατόμου, το αν λόγω ατόμου. Ευχαριστώ πολύ η εκπρόσωπος της ECR, η κυρία Ανδρέασεν. Δεν θέλετε. Όχι. Ο κύριος Δεγιό, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ δύσκολο να καταλήξουμε κάπου Δίκιο έχει ο κύριο Στάς, γιατί πολλές απαντήσεις δεν έχουμε λάβει, γιατί ε, η έρευνα δεν έχει τελειώσει. Έχουμε πάντως την εντύπωση ότι και οι αρχές της Μάλτας ε, δεν έχουν σκοπό να συνεχίσουν την έρευνα της ε, Όλαφ και επομένως δεν θα υπάρξουν διώξει κατά του κυρίου Νταλή. Αυτό προστίθεται, αυτή η υπόθεση προστίθεται σε άλλε υποθέσει όπου δεν υπήρξε συνέχεια σε επίπεδο κράτους μέλου των ερευνών τη. <clears throat> Όλαφ. Αυτή, ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολύ συχνά ε, αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Όλαφ ως ε, προστάτη των οικονομικών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέτε 43%, των αποτελεσμάτων της Όλαφ δεν ακολουθούνται από τις ε, χώρες μέλη. Είναι αλήθεια αυτό. Ευχαριστώ κύριο Κέσλερ. Κοιτάξτε, αυτή είναι μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια και δεν έχει ακόμα ε, ολοκληρωθεί. Έγινε και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού. Δεν ξέρω αν αυτό το στοιχείο, το στατιστικό του 43% ισχύει πραγματικά. Η διακύμανση είναι μεγάλη. Υπάρχουν χώρες με 3%, άλλες χώρες με 80%. Ε, νομίζω ότι είναι ένα θέμα πολιτικό, νομοθετικό ε, γιατί τα νομοθετικά πλαίσια που διέπουν τις απάτες διαφέρουν από χώρα σε χώρα Επίσης ε, όλα τα θέματα αυτά ξέρετε ότι ελέγχονται και από την οδηγία ΠΥΦΕ για την ε, ε, ποινική προστασία των οικονομικών δικαιωμάτων, συγγνώμη, συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, στην περίπτωση Νταλή, δεν υπάρχει έλλειψη ε, δίωξης, δεν θα πρέπει να προσμετρηθεί στο 33% γιατί ξεκίνησε διαδικασία και, ε, έχει, και συνεχίζεται ακόμα η ποινική διερεύνηση. Δεν θέλω να το αποκαλέσω επιτυχία, αλλά εδώ υπάρχει, ε, ε, έχει δοθεί συνέχεια στην ε, έρευνα της Όλαφ και ένας ανεξάρτητος δικαστής ασχολείται στην Μάλτα με το θέμα αυτό. Ε, υπήρξε μάλιστα και μία ε, προφυλάκηση όσον αφορά το ζήτημα ε, αυτό μεταξύ βεβαίως έχει ελευθερωθεί ο εν λόγω ε, κυρίως αλλά εν πάση περιπτώσει. Μια σύντομη συμπληρωματική ερώτηση. 43% αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο μας έχει ήδη δώσει και η Επιτροπή. Αν δεν είναι ορθό θα πρέπει να μας το πείτε. Απαντήστε μου απλά, ναι ή όχι. Η Όλαφ είναι διατεθειμένη να δεχθεί μια εξωτερική έρευνα ποιότητας για αυτό το 43%. Ένα λεπτό κύριε Κέσλερ. Βεβαίως και είμαστε διατεθειμένοι. Επίσης, έχουμε ξεκινήσει αυτόν τον διάλογο και έχουμε εντοπίσει εξωτερική έρευνα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στον επόμενο γύρο ερωτήσεων. Ελκ, όσον πια για ένα λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Κέσλερ, υπήρξατε πολιτικός, γνωρίζετε πολύ καλά τη λειτουργία της ε, δημοκρατίας. Ήσασταν βουλευτή στην Ιταλία από το 2001 στο 2006 και γνωρίζετε το ρόλο του Κοινοβουλίου όσον αφορά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας σε περιπτώσεις καταπολέμησης της απάτης. Εδώ βλέπετε ότι μεταξύ ημών και μελών αυτής της Επιτροπής δημιουργείται μια αντιπαράθεση. Το ερώτημα μου λοιπόν είναι, αν υπάρξει πρόταση μομφής, αν υπάρξει μια έκφραση δυσπιστίας, είστε διατεθειμένος να παρετηθείτε από Γενικός Διευθυντής της Όλαφ. Δύο λεπτά έχετε κύριε Κέσλερ. Ναι. νομίζω ότι θα υπάρξει αμφισβήτηση. Η απάντησή μου είναι όχι, όχι, όχι. Γιατί αν έκανα κάτι τέτοιο θα κατέστρεφα την ανεξαρτησία της Όλαφ. Θα εγκατέλειπα αυτή την ανεξαρτησία και δεν είναι ο ρόλος μου. Δεν προβλέπει κάτι τέτοιο ο κανονισμός της Όλαφ που ορίζει με μεγάλη σαφήνεια ότι σε αυτές τις διερευνήσεις, το ξεκίνημα, τη διεκπαιρέωση και το πέρας αυτών των ερευνών, η Όλαφ δεν θα πρέπει να δεχθεί καμία πίεση ή επιρροή από κανένα κράτος μέλος, κανένα θεσμικό όργανο. Δεν πρέπει να δεχθεί οδηγίες οι αιτήματα από κανένα θεσμικό όργανο. Αν έκανα λοιπόν κάτι τέτοιο, θα ήμουν αποτυχημένος ως προς την αποστολή μου για ανεξαρτησία. Δεν είναι δυνατόν να δεχτώ καμία πίεση, καμία εντολή από κανένα θεσμικό όργανο, κανένα πολιτικό φορέα. Συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Οντή. Μια παρατήρηση, δεν είναι ερώτηση κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί ένα τέτοιο λειτουργήμα χωρίς την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι σοσιαλιστές είναι η επόμενη ομάδα που θα κάνει ερώτηση. Η κυρία Γιάλα Σέντερ έχει ένα λεπτό. Ευχαριστώ. πλοκή κατάσταση. Πιστεύω ότι Όλαφ είναι κάπως αποδεπομπέος τράγος μιας απόφασης που ξεκινάει από πιο πάνω από τον πρόεδρο Μπαρόσο. Και για νομίζω ότι εκεί πρέπει να ζητήσουμε τη ρίζα της όλης υπόθεσης στην Κομισιόν. Κύριε Κέσλερ, και εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μια αντίφαση και σας είχα υποβάλει μια ερώτηση σας είχα πει αν η Όλαφ καταπολεμώντας ε, ε, το καπνό μήπως έχει πρόβλημα με τις πολυεθνικές ε, καπνού, μήπως έχει κάποια χρηματοδότηση στο πλαίσιο των... με τις πολυεθνικές. Και έλεγα ότι θα έπρεπε να ήταν κατεπήγον στην έρευνα η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων. Εσείς μου είχατε πει τότε ναι ότι υπάρχουν συμφωνίες και ένα μέρος της ε, χρηματοδότησης όλα εξαρτάται από την καταπολέμηση, τη θετική καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνού. Σε ό,τι αφορά επίσης ε, τις υποκλοπές, είπατε ότι ε, το να χρησιμοποιηθεί μια μαγνητοφωνημένη τηλεφωνική συνομιλία δεν είναι παράνομη, ε, στη χώρα μου είναι. Η δικαστές ε, δεν έλαβαν υπόψη ακόμη και σε υποθέσεις ε, με μαφιόζους και τρομοκράτες τηλεφωνικές συνομιλίες που είχαν υποκλαπεί. Χωρίς να το γνωρίζει δηλαδή ο εν λόγω. Θέλω να μου πείτε λοιπόν γιατί χρησιμοποιήσατε αυτή την κλίση και την άλλη ε, που κατεγράφει από την Όλαφ δεν τη χρησιμοποίησατε λέτε. τελικά τι γίνεται. Χωρίς να υπάρχει κανένα δικαστικό πλαίσιο μπορεί κανείς να είναι αντικείμενο υποκλοπής τηλεφωνικής. Γι' αυτό να πολύ. Σας ευχαριστώ. Έχετε δύο λεπτά κύριε Κέσλη. Οι συμφωνίες με τις ε, εταιρείε καπνού. Ουσιαστικά πρόκειται για δικαστικές, αν θέλετε, συμφωνίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτές οι συμφωνίες ακολούθησαν μια υπόθεση στις Ηνωμένε Πολιτείες και κατόπιν στην Ευρώπη κάποια κρατημέλη, όλα τα κρατημέλη, η Επιτροπή και οι εταιρείες, οι καπνοβιομηχανίες προχώρησαν σε αυτές τις συμφωνίες. Δεν ήταν η Όλαφ εμπλεκόμενη. Σαν αποτέλεσμα αυτών των συμφωνιών ουσιαστικά η Όλαφ δεν λαμβάνει απολύτως καμία χρηματοδότηση. Τα κράτη-μέλη ναι, η Επιτροπή ναι. Και τότε η, εταιρεία, η Επιτροπή συγγνώμη, Ελέγχου του Προπολογισμού είχε αναφερθεί σε αυτήν την χρηματοδότηση. Η Όλαφ δεν έχει καμία συμφωνία και δεν λαμβάνει καμία χρηματοδότηση από την καπνοβιομηχανία. Όσον αφορά την μαγνητοφώνηση αυτών των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων δεν το κάναμε σε καμία περίπτωση. Όσον αφορά τις τηλεφωνικές συνομιλίες ιδιωτικών προσώπων, σας είπα ότι δύο φορές έγινε αυτή η παρακολούθηση και η μαγνητοφώνηση, τη μία χωρίς να είμαστε παρόντες και τη μία μόνο χρησιμοποιήθηκε σαν αποδεικτικό στοιχείο στο δικαστήριο. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Αγιάλα Σέντερ, έχετε άλλη ερώτηση. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Σύντομα προς τον κύριο Κέσλερ. Όταν ξεκινά τις απαντήσεις, λέτε ότι ο Γενικός Διευθυντής δεν ήσασταν μεταξύ των ε, ανακριτών ή αυτών που ανέλαβαν την διέρευνηση της υπόθεσης, τέλος πάντων. Θα ήθελα να μας ε, ορίσετε το δικό σας ρόλο. Διότι πήγατε στη Μάλτα, είχατε συνεντεύξεις με κόσμο. Ε, ο ρόλος σας δεν είναι ρόλος ανακριτή ή τέλος πάντων ερευνώντος, τι ακριβώς είναι, πώς θα χαρακτηρίζετε το δικό σας ρόλο. Γιατί ακριβώς και με βάση αυτή τη πολύ δραστήρια συμμετοχή σα σε αυτή την έρευνα, είμαστε σε αυτή την κατάσταση για την Όλαφ, που έχουν προκύψει πολλά ερωτηματικά. Στο News Europe είδα και οι άλλοι, είδαμε ε, αλληλογραφία μεταξύ ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ ΣΑΝΚΟ και της Γενικής Γραμματείας σε σχέση με την ε, αναθεώρηση οδηγία και εκεί κάτι έπρεπε να είχατε καταλάβει, να είχε ηχήσει ως ένα γερμός. Απάντησε, να ξεκινήσω από το τέλος. Λέτε ότι υπήρξε μια ανταλλαγή αλλογραφίας η οποία βγήκε στο News Europe. Ναι, και εγώ τις ε, είδα, τις διάβασα και τη βάζω τελεία. Εμείς δεν έχουμε στο φακελό μας κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει κάτι, αλλά δεν είναι το θέμα που έχω εγώ, με το οποίο έχω εγώ ασχοληθεί. Οπότε, απλά σημειώνω αυτή την παρατήρηση για το δικό μου ρόλο. Εγώ είμαι ο Γενικός Διευθυντής της Όλαφ. Δυνάμει του κανονισμού, που σχεδόν ξέρω απ' έξω, Είμαι αυτός ο οποίος είμαι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή της έρευνας. Ανοίγω και κλείνω, σύμφωνα με τον κανονισμό, όλες τις έρευνες. Και ακριβώς πάντα σύμφωνα με τον κανονισμό, και δεν μπορώ καν να εκχωρήσω αλλού αυτή την αρμοδιότητα, είμαι αυτός ο οποίος πρέπει να δώσει έγκριση για όλες τις ε, έρευνες, τις πράξεις, ε, τις ερευνητικές που διεξάγονται από την όλα. Με μια συνέντευξη, οποιαδήποτε πρέπει να γίνει με πρώτερη δική μου γραπτή έγκριση. Το γράφει ο κανονισμός. Πρέπει να δώσω γραπτό στην εντολή εγώ. Άρα είμαι υπεύθυνο για οποιαδήποτε πράξη έρευνα. Είμαι υπεύθυνο για τη διεξαγωγή τη έρευνα, για το άνοιγμα και για το κλείσιμο τη έρευνα. Τώρα το αν αυτό με κάνει να είμαι ένας από τους δεν ξέρω, αλλά είμαι σίγουρα αυτός που τον τελευταίο λόγο. Και για τις συνεντεύξεις. Εάν ε, ένας ανακριτής ή ένας ερευνητής κάνει μια συνέντευξη, πρέπει να δείξει χαρτί που έχω υπογράψει εγώ, που του το επιτρέπει. Σε κάποιες συνεντεύξεις ε, που είχα εγώ εγκρίνει να γίνουν, συμμετείχα. Είμαι και ο τελευταίος υπεύθυνο πρώτα απ' όλα. Σε όλες δεν πήγα, αλλά σε κάποιες ήμουν παρόν. Μαζί με τους ερευνητές, τους ανακριτές. Ο εκπρόσωπος της Άλδε, όχι, των Πρασίνων, Μπάρτ. Λοιπόν, κύριε Κέσλερ, ας επανέλθουμε σε αυτήν την περίεργη εβδομάδα της 15ης Οκτωβρίου, στη διάρκεια της οποίας οι υπηρεσίε σας ε, μεταφέρουν, μεταβιβάζουν μάλλον το, το θέμα, το φάκελο στην ε, κυρία ε, Ντέιτζη. Και μετά από τρεις μέρες έχουμε μία ε, ε, ε, εν μέρη πληροφορείτε, μάλλον μερικώς πληροφορείτε την Επιτροπή Εποπτείας και λέτε τους έδωσα τρεις μέρες περιθώριο γιατί ήδη γνώριζαν το θέμα. Το ξέρατε όμως ότι υπήρχαν διαρροές στην κοινή γνώμη γιατί είχατε ήδη έρθει σε επαφή με τον πρόεδρο Μπαρόζο. Ξέρατε ότι ο πρόεδρος Μπαρόζο είχε ήδη συζητήσει με τον Επίτροπο Νταλή ο οποίος είχε παραιτηθεί. Είχατε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσετε πέντε μέρες ε, για την πληροφόρηση της Επιτροπής Εποπτείας γιατί ε, αν το είχατε κάνει θα είχαν, ε, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Θα είχε πέντε μέρες η Επιτροπή Εποπτείας να μελετήσει το θέμα. Ο ε, κύριος ε, Μπαρόζο θα είχε ζητήσει τη γνώμη της Επιτροπής Εποπτείας λοιπόν επί του θέματος αυτού και επομένως όλη αυτή η υπόθεση θα είχε αντιμετωπιστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια και με μεγαλύτερη ε, ταχύτητα. γιατί δεν ζητήσατε και από τον κύριο, από τον πρόεδρο Μπαρόζο να περιμένει πέντε μέρες μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Απάντηση. Κοιτάξτε, εγώ δεν είχα καμία επαφή με τον πρόεδρο Μπαρόζο πριν, κατά τη διάρκεια ή μετά την έρευνα. Καμία άμεση επαφή. Ε, ε, για να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα. Η Κάθριν Ντέι ήταν αυτή η οποία έδωσε αρχικά την πληροφόρηση στην ε, Όλαφ. Φαντάζομαι σαφώς μετά εκπροσωπώντας τον πρόεδρο Μπαρόζο και γι' αυτό ακριβώς εμείς δώσαμε ε, την τελική, το τελικό πόρισμα στην ε, κυρία Κάθριν Ντέι ε, και ήταν σαν να το δίναμε και στον πρόεδρο Μπαρόζο. Εμείς δεν είχαμε άμεση επαφή με τον πρόεδρο Μπαρόζο, καμία στιγμή σε καμία στιγμή, ούτε είχα καμία συμφωνία ή ουδήποτε είδους με τον πρόεδρο Μπαρόζο. Δεν ε, με εγκαλέσατε από αυτού, αλλά θα ήθελα να το διευκρινίσουμε παρόλα αυτά, έτσι ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε παρανόηση από αυτού. Σαφώς λοιπόν σας ε, απαντώ και αυτό φαίνεται άλλωστε και στα έγγραφα. Στείλαμε το φάκελο στην Κομισιόν και ταυτοχρόνως προετοιμάσαμε το φάκελο για την Επιτροπή Εποπτείας. Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να περιμένουμε ε, την γνωμοδότηση της Επιτροπής Εποπτείας ή ε, να στείλουμε πρώτα στην Επιτροπή Εποπτείας και μετά στα θεσμικά όργανα. Το κάνουμε διαρκώς, εκατό φορές το χρόνο, χωρίς να παραπονεθεί κανείς για παράβαση του κανονισμού. Απλώς πρέπει ε, να στείλουμε την πληροφόρηση στην Επιτροπή Εποπτείας πριν προωθήσουμε το φάκελο στη δικαιοσύνη. Και το κάναμε αυτό. Δεν θα μπορούσαμε ταυτόχρονα να στείλουμε δηλαδή το ζήτημα και στην Επιτροπή Εποπτείας και ε, στην, ε, στα δικαστήρια. Σύμφωνα με τον κανονισμό πρέπει πρώτα να στείλουμε την πληροφόρηση στην Επιτροπή Εποπτείας και μετά στα δικαστήρια. Ε, λέτε ότι στείλαμε μερική πληροφόρηση στην Επιτροπή Εποπτείας. Εν μέρει ισχύει. Στείλαμε στην Επιτροπή την έκθεση και τις συνεντεύξεις. Δεν στείλαμε στην Κομισιόν όλο το φάκελο, δεν ήθιστε, δεν αποτελεί συνήθη πρακτική και δεν το κάνουμε και τούτη τη φορά. Αυτό που στείλαμε στην Επιτροπή Εποπτείας όμως είναι ακριβώς οτιδήποτε ε, γράφτηκε, γράφεται στην ε, συμφωνία εργασίας και συνεργασίας μαζί τους. Ε, και αυτό βασίζεται σε ε, σε νομικά δεσμευτική γνωμοδότηση ε, του ε, επόπτη δεδομένων. Προβλέπετε λοιπόν ότι πρέπει να δοθεί μία έκθεση η οποία θα είναι σύντομη και η οποία δεν θα αναφέρεται ε, σε συγκεκριμένα ονόματα. Αυτή είναι η μερική πληροφόρηση. Είμαστε υποχρεωμένοι να στείλουμε αυτή τη μερική πληροφόρηση. Όμως εκείνη, αυτό που συνέβη είναι ότι εκείνοι μόλις έλαβαν την πληροφόρηση μας ζήτησαν να έχουν πλήρη πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία και ζήτησαν ένα μήνα, όχι δύο μέρες, ένα μήνα. Και δεν μας ζήτησαν να περιμένουμε, ποτέ δεν συμβαίνει αυτό. Ποτέ δεν μας ζητήθηκε να περιμένουμε και ποτέ δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Επομένως, απέκτησαν πλήρη πρόσβαση στο φάκελο πριν καν στείλουμε εμείς το θέμα στα δικαστήρια. Η ECR έχει τη δυνατότητα να κάνει ερώτηση. Κυρία Ανδρέασεν. Όχι. Ολοκληρώσαμε λοιπόν αυτό το γύρο ερωτήσεων. Θα δώσω τώρα το λόγο πάλι στο ΕΛΚ. Κυρία Γκρέσλε, ευχαριστώ πολύ. Είναι ενδιαφέρον, κύριε Κέσλερ, να ακούσει κανείς τη συζήτησή σας. Επαναλαμβάνετε ότι όλα είναι νόμιμα μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο ενώπιον των δικαστηρίων. Δηλαδή, εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω κάποια πράγματα όταν μου το ορίσει το δικαστήριο. Κοιτάξτε, ίσως θα πρέπει να ξαναδείτε λίγο αυτά που πρέπει να κάνετε, γιατί θεωρώ πραγματικά ότι δεν είναι αυτό μήνυμα για να στείλουμε προς τα έξω. Ότι μέχρι δηλαδή να αποδειχθεί η παρανομία είμαστε νόμιμοι. Δηλαδή χωρίς απόφαση δικαστηρίου θα συνεχίσετε αυτές τις πρακτικές, τις οποίες χαρακτηρίζετε νόμιμες. Αυτές οι τηλεφωνικές συνομιλίες με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα. Επίσης, το γεγονός ότι κάποιος παρακολουθεί μία τηλεφωνική συνδιάλεξη και την μαγνητοφωνή χωρίς ένας από τους δύο συνομιλούντες να το γνωρίζει. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Κύριε Κέσλερ, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Όσον αφορά την νομιμότητα, κοιτάξτε, οτιδήποτε είναι παράνομο, είναι, ε, είναι παράνομο οτιδήποτε είναι κατά του νόμου. Σε πολλές φορές όμως υπάρχουν διαφορετικές ερμηνείες, διαφορετικές γνώμες για το τι είναι νόμιμο και τι δεν είναι νόμιμο. Γι' αυτό υπάρχουν τα δικαστήρια. Δεν αποφασίζω εγώ ή εσείς, αποφασίζουν τα δικαστήρια και μια ολόκληρη σειρά διαδικασιών έτσι ώστε να καθοριστεί αν κάτι είναι σύμφωνο με τον νόμο ή παράνομο. Για τις α, τηλεφωνικές συνομιλίες επαναλαμβάνω αυτό που ήδη σας είπα. Και δεν μπορώ να πω τίποτα παραπάνω για το τι συνέβη. Όπως σας είπα, συνέβη δύο φορές κατά την άποψή μας σε πλήρη νομιμότητα, μία πριν την έρευνα και μία κατά τη διάρκεια της έρευνας από ένα ιδιώτη και αν διαβάσετε την έκθεση της Επιτροπής Εποπτείας, όλα αυτά αναφέρονται. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα παραπάνω. Αν είναι παράνομο, κάποιος θα πρέπει να το αποφασίσει. Εμείς όμως επαναλαμβάνουμε ότι δεν κάναμε απολύτως τίποτα. Εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε σε καμία τηλεφωνική συνδιάλεξη. Δεν χρησιμοποίησαμε λοιπόν κανένα μέσο, καμία εξουσία για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκρέσλε. Όλα αυτά ήταν στα κτίρια της Όλαφ, παρουσία λειτουργών της Όλαφ, τι να σας πω. Εδώ υπάρχει μια σημαντική παρανόηση όσον αφορά την ανεξαρτησία της Όλαφ. Εμείς θέλουμε να υπάρχει ανεξαρτησία και ανεξάρτητη έρευνα. Απλώς θέλουμε να υπάρχει και δυνατότητα κατόπιν αξιολόγησης ελέγχου από μέρους μας και πραγματικά σε καμία περίπτωση δεν λειτουργείται σαν ε, ελεύθερος φορέας χωρίς κανένα έλεγχο ποτέ. Τώρα, το θέμα είναι αν πρόκειται για απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής ναι ή όχι. Επίσης το θέμα του καταστατικού και του άρθρου 220 Γνωρίζετε το άρθρο αυτό και τι έχετε να πείτε για την ερμηνεία του. Κύριε Κέσλερ, έχετε ένα λεπτό, λέει ο πρόεδρος. Βεβαίως και το γνωρίζω. Η σοσιαλιστική ομάδα έχει τη δυνατότητα να κάνει άλλη μια ερώτηση. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο εκ μέρους των σοσιαλιστών. Όχι. Η, ΕΛΚ, λοιπόν, η ομάδα του ΕΛΚ λοιπόν έχει τελικά άλλη μια ερώτηση κυρία Γκρέσλε. Θα επανέλθω στο θέμα του ρόλου που παίζουν διάφοροι συνεργάτες της Όλαφ και παραδείγματος χάρη ενώπιν της διαδικασίας με το ελεκτικό συνέδριο αλλά και το θέμα με τους μάρτυρες κατηγορίας. Γιατί χρησιμοποίησε η όλα αυτές τις μεθόδους. Εδώ ουσιαστικά πρόκειται για θέμα αρχής. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Όλαφ χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία με αυτόν τον τρόπο. Και εδώ αναφέρομαι στην ερώτηση 35C και D και περιμένω μία απάντηση. Και πάλι τα συζητήσαμε αυτά. Και συγγνώμη, συζητώνται ενώπιον του δικαστηρίου αυτές τις μέρες. Είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται. Τι λεπτομέρειες να σας δώσω χωρίς να παρέμβω στη δικαστική διαδικασία. Αναφέρεστε σε κάτι το οποίο σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί χρήση ή κατάχρηση εξουσίας. Τι να σας πω, είναι σαν κάποιος να πηγαίνει κάπου σε μια συγκεκριμένη διεύθυνση και να βλέπει παραδείγματο χάλιν στο κουδούνι στην πόρτα τι όνομα υπάρχει. Αυτό μπορεί να συμβεί. Πηγαίνει ένας συνεργάτης της Όλαφ για να διαπιστώσει αν στο κουδούνι της πόρτας υπάρχει ένα συγκεκριμένο όνομα. Μα τι κατάχρηση εξουσίας ε, μπορεί να αποτελέσει αυτό. Είναι μια απλή δραστηριότητα την οποία μπορεί ο κάθε Ευρωπαίος πολίτης ε, να αναλάβει. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκρέσλα, έχετε ένα λεπτό. Μα εδώ δεν μιλάμε για κανονικούς πολίτες, μιλάμε για την Όλαφ που διεκπεραιώνει έρευνες. Και εδώ θα πρέπει σαφώς να τηρούνται οι εγγυήσει και το κράτος δικαίου. Γιατί όπως ξέρετε η Όλαφ χρησιμοποιεί διάφορες ε, ταυτότητες για να μην διαπιστωθεί από τους ε, μάρτυρες ε, ποιοι ακριβώς είναι. Μα δεν γνωρίζω αυτό που λέτε, λέει ο κύριος Κέσλερ. Σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις δεν συνέβη κάτι τέτοιο. Δεν βλέπω κάποιον να ζητάει το λόγο, γι' αυτό και θα θεωρήσω ότι τελείωσε η σειρά των ερωτήσεων. Εγώ έχω μία συμπληρωματική ερώτηση, κύριε Κέσλερ, σαν πρόεδρος. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα τα αποτελέσματα της ε, έρευνας αυτής της Όλαφ να χρησιμοποιηθούν σαν πολιτικό εργαλείο και τι μέτρα θέλετε να ληφθούν στο μέλλον έτσι ώστε να μην υπάρχει τέτοιου είδους δυνατότητα κατάχρησης. Τώρα είμαι σε θέση να σας ε, κάνω τις υποδείξεις που μου ζητάτε. Όλοι άλλωστε, <clears throat> και τα θεσμικά και όχι μόνο όλα θα πρέπει να λαμβάνουν ενδεχομένω αυτές τις υποδείξεις γιατί για τη θεωρητική περίπτωση που αναφέρεται μπορεί και από πολιτικούς να χρησιμοποιηθούν αυτά τα μέσα. Η πρώτη προφύλαξη λοιπόν που χρησιμοποιούμε και εμείς και χρησιμοποιήσαμε είναι να μην οφείλουμε να διαρρεύσει κάτι. Και νομίζω το καταφέραμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Σας λέω ότι αυτή ήταν η βασική μου με τους πέντε μήνες αυτούς επειδή υπήρχε μεγάλος κίνδυνος διαρροών. Για να μην ε, δημοσιοποιηθούν οι πληροφορίες λοιπόν και μετά ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν από κάποιον για πολιτικούς λόγους πριν γίνουν οι διευκρινήσεις οι απαραίτητες εγώ υποχρεούμε από τον νόμο, από τον κανονισμό να στείλω τα αποτελέσματα. στον ενδιαφερόμενο οργανισμό και στην προηγούμενη περίπτωση και στις δικαστικές αρχές. Το πράξαμε, αλλά με εμπιστευτικότητα. Έπειτα, συνήθισαν πολιτικά συμπεράσματα. Αυτά φαντάζομαι δεν μπορώ να είναι να παραμείνουν μυστικά και αυτός και συνέβη. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες ε, υποδείξεις, δεν ξέρω. Μήπως δεν πρέπει να στέλνονται, για παράδειγμα, τα αποτελέσματα στα δημιουργικά όργανα ή στο οικείο, στο ενδιαφερόμενο. Εγώ νομίζω ότι το ενδιαφερόμενο όργανο πρέπει να ξέρει τα αποτελέσματα της έρευνας. Πρέπει όμως να λάβει ανεξάρτητα τις αποφάσεις του και με δική του ευθύνη. Σας ευχαριστώ πολύ. Η ερώτησή μου προκάλεσε αντιδράσεις βλέπω. Κυρία Γκρέσλε, εγώ θα ήθελα να ενημερώσω το Γενικό Διευθυντή ότι το Σεπτέμβριο Μίλησα με δύο εκπροσώπους της αυτοκινητοβιομηχανίας που αναφέρθηκε ακριβώς στις ε, περιπτώσεις επιτρόπων ε, που αντιμετωπίζουν αυτές τις διαδικασίες. Πρόεδρος, άλλες παρεμβάσεις δεν βλέπω κανέναν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Κέσλερ, ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής. Νομίζω ότι η διαδικασία που επιλέξαμε ήταν ε, επιτυχής γιατί μπορέσαμε να ανταλλάξουμε απόψεις. Ναι, θα σας δώσω το λόγο, αλλά θα ήθελα να διακόψω για λίγα λεπτά τη συνεδρίαση και να ξαναρχίσουμε στις 12 παρατέταρτο. Ναι, εγώ θα ήθελα να ζητήσω η Κάθριν Ντέι και η κυρία Κότσι να έρθουν εδώ. Ναι, την Γενική Γραμματέα Ντέι και την κυρία Τέστορη Κότσι. Σύντομα κύριε Πρόεδρε, από τη στιγμή που ο Γενικός Διευθυντής αρνείται να παραιτηθεί σε περίπτωση που το κοινό Κοινοβούλιο καταθέσει πρόταση πιστείας ή μόφης εναντίον του, πιστεύω ότι πρέπει να ζητήσουμε μια νομική ονομάτευση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πρακτικά, πώς μπορούμε να καλέσουμε ε, από τα καθήκοντά του τον ε, Γενικό Διευθυντή. Αν θεωρούμε ότι πλέον δεν μπορεί να είναι ηγείται της Όλαφ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Μούλντερ. Εγώ στηρίζω το της κυρίας Κρέσλερ για την ακρόαση αυτών των δύο προσώπων εδώ στην Επιτροπή. Ναι, άκουσα λοιπόν να καλέσουμε την Γενική Γραμματέα της Επιτροπής. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις μας. Θα δούμε βεβαίως τι θα μας πει και ο Επίτροπος Σέμετα. Τώρα, το θέμα που έθιξε ο Ζωμπιέγο Οντί θα το ελέγξει η γραμματεία και θα σας ενημερώσουμε. Ολοκληρώσαμε με αυτό το σημείο, θα διακόψουμε για ένα τέταρτο και θα συνεχίσουμε την κανονική μας συνεδρία, την τακτική μας συνεδρίαση στις 11.45. Ε, Uh, Sigmantas, uh, would you be ready to... Είστε έτοιμος, συνάδελφε Σιγμάντας. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf wieder ein... Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, ξαναρχίζουμε τις εργασίες μας. Ευχαριστούμε πολύ για την ε, ε, συνεργασία και την κατανόηση νομίζω ότι μας άξιζε αυτή η διακοπή. Έχουμε το σημείο 19, ειδική έκθεση 21-2012 με θέμα την αποδοτικότητα των επενδύσεων που αποσκοπούν στην ενεργειακή αποδοτικότητα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Πήρε τη θέση του σημείου 13. Ο κύριος ε, ε, Μπαλσίτης ε, είναι ο εισηγητής και εκπρόσωπος του ελεγκτικού συνεδρίου ο κύριος Χάρναντ Βέγκερ Μπράουερ. Κύριε Μπαλσίτη παρακαλώ έχετε το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω το ελεγκτικό συνέδριο και τον εκπρόσωπό του που ε, μας έδωσε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, έγγραφο που αφορά ε, τρεις χώρες ε, στις οποίες ε, δόθηκαν τα μεγαλύτερα κονδύλια ε, και τα οποία αφορούσαν την ενεργειακή αποδοτικότητα και την ανακαίνιση. Τα αποτελέσματα δεν μας ικανοποιούν. Πρώτα απ' όλα είδαμε ότι δεν υπήρξε σύστημα ελέγχου ή εποπτείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν δώσει τα κονδύλια αυτά δεν έδωσε κριτήρια ή απαιτήσει Αναφερόμαστε εδώ στην περίοδο 2000-2006 ε, και αυτό συνδέεται με το δημοσιονομικό πλαίσιο ε, το σχετικό. Βεβαίως δεν μπορούμε να επανέλθουμε, να αλλάξουμε το παρελθόν. Να πούμε πάντως ότι σε μερικές χώρες μέλη ε, η η αποδοτικότητα αυτών των σχεδίων αφορά μία περίοδο 50 ετή και μερικές φορές 100 ετή. Το ελεγκτικό συνέδριο συστήνει να, συνδέονται, να συνδέεται το Ταμείο Συνοχής με καλή αξιολόγηση των αναγκών, ε, με την εποπτεία της χρήσης ε, των κονδυλίων βάσει συγκρίσιμων ε, κριτηρίων και επίσης κυρίως την χρήση τέτοιων κριτηρίων. Πράγμα πάρα πολύ σημαντικό εάν θέλουμε πραγματικά να καταφέρουμε να ορίσουμε τα καλύτερα ποσοστά ε, απόδοσης των επενδύσεων. Ε, γιατί ε, αυτά τα ζητήματα θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην κατανομή των κονδυλίων. Έχουμε σήμερα εκπρόσωπο και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Κομισιόν. Ε, πρέπει να συμφωνήσουμε με το γεγονός ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για όλα τα projects και επομένως θα πρέπει να καθοριστούν εκ των προτέρων ε, και τα κριτήρια και οι υποχρεώσεις και οι δείκτες βάσει των οποίων μπορεί να γίνει αξιολόγηση της αποδοτικότητας ε, των επενδύσεων. Συμφωνούμε λοιπόν όλοι ότι πρέπει να καθοριστούν και κόστη ανά ενεργειακή κατηγορία. 20% των κονδυλίων θα πρέπει ε, να ε, δοθούν στην βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. έτσι ώστε να επιτευχθούν οι 20 στόχοι της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ε, εδώ πρέπει να δούμε επίσης και την εμπειρία κάποιων κρατών μελών. Ας πούμε το παράδειγμα της Γαλλίας να πάρω. Ε, στην ανακαίνιση ενός ε, Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι έχουμε 500 τετραγωνικά. Ε, εδώ μπορούμε ε, για να επιτύχουμε τους στόχους θα πρέπει να έχουμε εξοικονόμηση τουλάχιστον 30% ε, της ενέργειας. Μόνο με τον τρόπο αυτό θα χρησιμοποιείται αποτελεσματικά το χρήμα του Ευρωπαίου φορολογούμενου. Κοιτάξτε, τα ζητήματα αυτά είναι ιδιαίτερα περίπλοκα και θα πρέπει να επανέλθουμε σε αυτά και στο μέλλον, διότι σε κάθε project υπάρχουν ε, ε, διαφορετικές φάσεις Τέσσερις-πέντε φάσεις ανάλογα με τον όγκο του, του project και ανάλογα ε, με την αποδοτικότητα που θέλουμε να επιτύχουμε. Επομένως ε, κάθε project θα πρέπει να, είναι, να μελετάτε ξεχωριστά ε, και οι προθεσμίες να είναι διαφορετικές αναπερίπτωση. Το ελεγκτικό συνέδριο υπεγράμισε ήδη το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχει και ο έλεγχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αρμόδια Γενική Διεύθυνση εξεφράστη, εξέφρασε τη γνωμοδότησή της και είπε ότι η Κομισιόν δεν μπορεί να είναι ε, υπεύθυνη για όλα τα προγράμματα ε, και για όλα τα σχέδια ε, παρόλα αυτά πρέπει να προβλεφθεί ένα ενιαίο σύστημα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει του οποίου ε, να είμαστε σε θέση να κατανοήσουμε αν τα κράτη-μέλη κατάφεραν να επιτύχουν τον στόχο ενεργειακής απόδοσης που είχαν θέσει εξ αρχής. δε, πρέπει να γίνουν όλα αυτά έτσι ώστε να μην πούμε μετά από μερικά χρόνια ότι δυστυχώς δεν επιτύχαμε τους στόχους παρότι τα κονδύλια έχουν ε, ε, χρησιμοποιηθεί. Τελειώνοντας να ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά και το Ελεγκτικό Συνέδριο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατανόησή τους. Νομίζω ότι στο έγγραφο εργασίας μου θα αναφερθώ ε, σε αυτές τις ε, αρχές οι οποίες ε, θα είναι χρήσιμες και για το μέλλον κατά την άποψή μου. Και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιασδήποτε ερωτήσεις αλλά και να απαντήσω στις συστάσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Βέγκεμπαουερ από το ελεγκτικό συνέδριο. Α, ο κύριος Βαλσίτης. Ευχαριστώ. Ο εισηγητής ε, ήδη έχει πάρει κάποια στοιχεία από τις συστάσεις του ελεγκτικού ε, συνεδρίου και είμαστε πολύ ευτυχείς γιατί θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε κοινή προσέγγιση από εδώ και πέρα. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Επίσης είδαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντέδρασε με πολύ θετικό τρόπο σε αυτά που συμπεριλάβαμε στην έκθεσή μας και αυτός είναι και ο σκοπός μιας έκθεσης του ελεγκτικού ε, συνεδρίου, δηλαδή να βελτιωθεί η κατάσταση ε, στο μέλλον. Και θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ε, στάση. Θα ήθελα παρόλα αυτά πολύ σύντομα να σας παρουσιάσω τις σημαντικές πτυχές αυτής της έκθεσης για να ενημερωθείτε κυρίως για ποια είναι τα σημεία στα οποία θέλουμε να επικεντρωθούμε. Τα κύρια στοιχεία αυτής της πρότασης που αφορά τα πέντε δισεκατομμύρια ευρώ για την πολιτική συνοχής και τη χρηματοδότηση, τα προγράμματα τα οποία έχουν επιλεγεί. Πρόκειται για την περίοδο 2014-2020 και εδώ αναφερόμαστε σε ένα ποσό που ξεπερνά την αρχική χρηματοδότηση. Σκοπός μας είναι μέχρι το 2020 να μειωθούν οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα κατά 20%. Εδώ ουσιαστικά πρόκειται για μια παράλληλη μείωση του κόστους στον τομέα της ενέργειας και την ίδια ώρα μια σημαντική εξοικονόμηση στον ίδιο τομέα. Και βεβαίως αυτό για να υπάρχουν πιο αποτελεσματικές ε, εγκαταστάσεις και εξοπλισμοί στα παράθυρα, παραδείγματος χάρη, και μέχρι τώρα ξέρουμε ότι χρησιμοποιήθηκαν κατά 20% τα κονδύλια αυτά όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας για μεγάλα προγράμματα επενδύσεων. Ένα σχέδιο, ένα πρόγραμμα στο οποίο επενδύθηκαν σε πολλούς τομείς το συνολικό κόστος λοιπόν αυτών των επενδύσεων δεν ήταν αποκλειστικά και μόνο στοχευμένο στην εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και στην ανακαίνιση, στην διακόσμηση. Όλα αυτά βεβαίως είναι πολύ αξιόλογα, δεν είναι όμως σε καμία περίπτωση σκοπός αυτού του μέτρου. Το Ευρωπαϊκό λοιπόν Ελεκτικό Συνέδριο έχει ελέγξει όλες αυτές τις επενδύσεις. Πρόκειται για χρηματοδότηση από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ταμεία για την περίοδο 2007-2013 στη Λιθουανία, Τσεχία και Ιταλία. Μέχρι το τέλος του 2011, 1,2 δις είχαν διατεθεί για προγράμματα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης Επιλέξαμε και κάποια προγράμματα τα οποία ελέγξαμε μέχρι το 2013. Τέσσερα προγράμματα τα οποία ελέγξαμε και συγκρίναμε με τις προβλεπόμενες δαπάνες για το 2014-2020. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι να δούμε κατά πόσον έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι για την εξοικονόμηση ενέργειας, χωρίς βεβαίως να συμπεριληφθούν και άλλες δαπάνες. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτών των προγραμμάτων. Τα προγράμματα τα οποία ελέγχθηκαν, ελέγχθηκαν ανατομέα, αναπεριφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες μεθόδους αξιολόγησης και εκτίμησης. Όσον αφορά την εκτίμηση του κόστους εξοικονόμησης και απόδοσης της ενέργειας, λάβαμε υπόψη μας τα μέτρα που ελήφθηκαν και πολύ θετικά παραδείγματα πρότυπα θα έλεγα είναι για μας η Δανία και το Βέλγιο. Με μία περίοδο πενταετή στη Δανία και μεγάλη εξοικονόμηση και απόδοση ενέργειας, αντίθετα στο Βέλγιο είδαμε ότι για μία επταετή περίοδο που ελέγχθηκε διαπιστώσαμε ότι η περίοδος υλοποίηση τελικά ήταν τριετής, κάτι το πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Για την Τσεχία είδαμε ότι ο χρόνος για την απόσβεση των επενδύσεων και για τις περιόδους και τα προγράμματα που ελέξαμε φτάνει από 28 έως 61 έτη για την Ιταλία. Επίσης τα αποτελέσματα ήταν ε, λιγότερο ενθαρρυντικά όσον αφορά τώρα την Τσεχία. Είδαμε ότι η περίοδος ε, για την απόσβεση των επενδύσεων ξεπερνάει τα 96 χρόνια σε κάποιες περιπτώσεις. Πρόκειται για πάρα πολύ ε, μεγάλες περιόδους για την απόσβεση. Όσον αφορά τις διάφορες ε, περιόδους που ελέγξαμε και τις ε, αν θέλετε δευτερεύουσες συνέπειες που είναι πέρα δηλαδή από την απόδοση την ενεργειακή ή άλλοι τομείς που βελτιώθηκαν. Για την Ιταλία δεν έχουμε τελικά αποτελέσματα, για την Λιθουανία ελέγξαμε δύο συγκεκριμένα προγράμματα, για την Τσεχία Ελέξαμε κτίρια και αξιολογήσαμε την ενεργειακή τους απόδοση. Οι ελεγκτές, οι επιθεωρητές επέλεξαν μία μέθοδο αξιολόγησης η οποία ενδεχομένως δεν ήταν η πιο οικονομική αλλά είχε τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την απόδοση την ενεργειακή ελέγξαμε δηλαδή την μόνωση ε, όσον αφορά τα πατώματα, τα παράθυρα, τις πόρτες. Επίσης ελήφθησαν υπόψη και η βελτιώση στον τομέα της ασφάλειας, κάτι που ήταν απλώς μια δευτερεύουσα συνέπεια. Επίσης στην Τσεχία κοιτάξαμε και τις ε, πραγματικές επιθεωρήσεις των αποτελεσμάτων, κάτι που δεν έγινε στις άλλες χώρες, γιατί στις άλλες χώρες οι ε, επιθεωρήσεις έγιναν βάσει των στοιχείων που μας παρήχαν. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κοιτάξουμε και τον εξοπλισμό αλλά και τα κτίρια. Πρέπει να σας πω ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν μια διάρκεια ε, για την απόσβεση των επενδύσεων πενταετίας έως, ε, από 5 δηλαδή έως 10 χρόνια. Αυτό είναι κάτι που οδήγησε σε μια χρησιμοποίηση των διατηθέμενων κονδυλίων της τάξης του 10%. Η διάρκεια της απόσβεσης ξεπέρασε τα 46 χρόνια στην Τσεχία, στην Ιταλία Πρέπει να σας πω ότι η περίοδος ήταν λιγότερο ε, μεγάλη αλλά πολύ σημαντική κατά την άποψή μας, 146 χρόνια για τη Λιθουανία. Πρέπει πραγματικά αυτά τα μέτρα για την εξοικονόμηση και της ενέργειας και την καλύτερη απόδοση να ειδωθούν σε σχέση με τα γενικότερα μέτρα και όχι μόνο κοιτώντας την απόδοση της ενέργειας. Αυτό είναι κάτι που σε καμία περίπτωση βεβαίως δεν μπορεί να εξεταστεί ανεξάρτητα από τις ε, υπόλοιπες συνέπειες όσον αφορά το συγκεκριμένο κόστος της χρηματοδότησης αναγκαστήκαμε να απομονώσουμε την περίοδο απόσβεσης που όπως σας είπα πολλές φορές φτάνει και τα 50 χρόνια. Το θέμα τώρα του στόχου για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα του 2020 κατά 20%. Αυτό βεβαίως από τη στιγμή που τα 17 δισεκατομμύρια που έχουν προβλεφθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διατεθούν στοχευμένα. Σε αυτή την περίπτωση πιστεύουμε ότι μπορούμε να μην ξεπεράσουμε το 10% και να μην φτάσουμε ποτέ στο 20% και αυτό βεβαίως από τη στιγμή που η κατανομή των κονδυλίων θα γίνει με τον προβλεπόμενο τρόπο. Τα αποτελέσματα τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πραγματικά ότι όσον αφορά την ανάλυση των αναγκών, όσον αφορά τις δυνατότητες εξοικονόμησης, οι στόχοι και η αξιολόγηση αυτών των μεθόδων και οι πιο οικονομικές μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν. Μπορέσαμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα βάσει συγκεκριμένων δικτών και συμπεριλαμβάνοντας όλους τους συντελεστές όσον αφορά την συνιστόσα του κόστους και βεβαίως την περίοδο απόσβεσης βάσει των δικτών που είχαν προκαθοριστεί. Οι εθνικές αρχές είναι αυτές που έχουν συλλέξει όλα αυτά τα στοιχεία και φυσικά η αξιολόγηση και ανάλυση έγινε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πολύ σημαντικό εδώ να ξαναδούμε την περίοδο απόσβεσης έτσι ώστε να επιλεγούν για το μέλλον οι πιο ε, οικονομικές και αποδοτικές λύσεις. Στο μέλλον επίσης θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε τα κριτήρια για να επιλεγούν τα προγράμματα που είναι τα πιο οικονομικά και αυτά που έχουν τα κατάλληλα αποτελέσματα όσον αφορά την απόδοση της ενέργειας. Συμπερασματικά θα ήθελα να συμπληρώσω ότι θα πρέπει εδώ να στηρίξουμε διάφορα μέτρα τα οποία έχουν αποδείξει την απόδοσή τους και όσον αφορά άλλους παράγοντες όπως την ανάπτυξη, την περιφερειακή, κάτι που εμπεριέχεται σαν συντελεστή στα διάφορα προγράμματα θα πρέπει ίσως να επιλέξουμε και άλλους τρόπους χρηματοδότησης και άλλες πηγές χρηματοδότησης. Σας ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Βογγενμπάου για την έκθεσή σας. Πριν δώσω το λόγο στην Επιτροπή, θα ήθελα να ρωτήσω τα μέλη της Επιτροπής μας αν θέλουν να πάρουν το λόγο. Δεν βλέπω κανένα ζητάει το λόγο. Η Επιτροπή λοιπόν. Uh, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και τον ε, κύριο Βουλευτή για την έκθεσή του, καθώς επίσης και τον εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Θεωρούμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η έκθεση αυτή είναι έγκαιρη, έρχεται τη σωστή στιγμή και ε, είναι πολύ θετική. Τέσσερις σκέψεις θα εκφράσω και μετά μια πολύ σύντομη εξήγηση σχετικά με το τι προτιθέμεθα να κάνουμε, έτσι ώστε να συμμορφωθούμε προς τις ε, υποδείξεις της έκθεσης. Το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να είναι το εξή. Στην προγραμματική περίοδο 2000-2006 οι 3 εκατομμύρια ευρώ δαπανήθηκαν για την ενεργειακή αποδοτικότητα, ε, πολλαπλασιαζόμενο από επί 15 ε, στην επόμενη προγραμματική περίοδο 2007 με 2014. Τεράστια αύξηση σε μικρή χρονική ε, περίοδο. γιατί η ενεργειακή αποδοτικότητα ήταν στόχος της ε, πολιτικής συνοχής. Τέσσερις σκέψεις λοιπόν όσον αφορά τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο της εκθέσεως του Ελεκτικού συνεδρίου. Πρώτον, πρέπει να αναγνωριστεί γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε σωστές μετρήσεις της ίδιας της πολιτικής. Πρέπει να υποθεί λοιπόν ότι η πολιτική μας εντάσσεται στην ε, γενικότερη πολιτική για την οικονομική ε, απόδοση. Δεν είναι τομιακή πολιτική. Να σας το εξηγήσω. Όταν ε, οικοδομούμε ας πούμε ε, σχολείο σε ε, μια φτωχή γειτονιά, ο αντίκτυπος είναι κοινωνικός και οικονομικός και θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης και η ενεργειακή αποδοτικότητα, αυτού του, η ενεργειακή αποδοτικότητα του ε, τμήματος, του σχολείου είναι ένα τμήμα του συνολικού προγράμματος. Ένα άλλο παράδειγμα. Όσον αφορά και το παράδειγμα της ε, Γαλλίας. 200 εκατομμύρια ευρώ στην προγραμματική περίοδο αυτή και η μόχλευση αφορούσε 1,2 δις ε, ε, επιπλέον χρηματοδότησης ε, κοινωνικής και περιφερειακής όσον αφορά την κοινωνική στέγαση, ιδωμένη και από την πλευρά της ενεργειακής αποδοτικότητας. 60.000 οικογένειες βοηθήθηκαν να ζήσουν καλύτερα και έτσι περαιτέρω δημιουργήθηκαν 16.000 θέσεις εργασίας επιτόπου γιατί θέλουμε να μιλήσουμε και για παραγωγικότητα και για ανάπτυξη. Η κατάσταση είναι η εξή. Ε, αυτή τη στιγμή υπάρχει κοινή διαχείριση. Να σας υπενθυμίσω ότι εμείς είμαστε όμως υπεύθυνοι για, την, την, ε, τον προϋπολογισμό. Τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για τον καθορισμό κριτηρίων επιλεξιμότητας ε, των προγραμμάτων, ε, είναι υπεύθυνη για την επιλογή των προγραμμάτων και τα κράτη-μέλη επίσης είναι ε, υπεύθυνα να το κάνουν, έχουν την ευθύνη δηλαδή να κάνουν κάτι τέτοιο βάσει το, της επιλογής των καλύτερων και πλέον συμφερουσών ε, διαδικασιών, προσφορών κτλ. Η Κομισιόν είναι υπεύθυνη όσον αφορά τα προγράμματα μονάχα ε, για την απόφαση επί των ε, μεγαλύτερων σχεδίων, των major projects. Επ' αυτού έχουμε μία ανάλυση κόστους-οφέλους πάρα πολύ προχωρημένη, την οποία δίνουμε και στα κράτη-μέλη. Για τούτη την προγραμματική περίοδο ε, η ε, Κομισιόν παίρνει απευθείας απόφαση για 700 major projects. Και εκεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει σε βάθος την κατάσταση όσον αφορά τη σχέση ωφέλους Δεν νομίζω ότι στο δείγμα που ελέγχθηκε υπήρχε ε, κάποιο major project. Όσον αφορά τώρα τις περιόδους αποπληρωμής και επίσης πώς αυτό σχετίζεται με το σκέλος της ενεργειακής αποδοτικότητας στην ανάλυση αυτή ε, υπό το φως των ευρυτέρων στόχων. Ε, ο χρόνος απόσβεσης διαφέρει βεβαίως και σχετίζεται με τον τρόπο με τον οποίο καθορίζει κανείς την εξοικονόμηση η οποία έχει, ε, έχει προκύψει σε 18 από τα 24 προγράμματα ε, αναφέρεται ότι δεν μπορεί αυτή η αξιοοικονόμηση να μετρηθεί. Με αυτούς τους όρους βεβαίως δύσκολα μπορεί κανείς να καθορίσει τις περιόδους απόσβεσης. Μπορεί κανείς να μιλήσει για 150 χρόνια. Ωραία, αυτό είναι θεαματικό, συνέβη σε, μία, σε ένα ε, project μόνο, αλλά οπωσδήποτε δεν αποτελεί κοινό μέτρο και δεν ισχύει για όλα τα project. Οι συγκρίσεις όσον αφορά την περίοδο απόσβεσης είναι εξαιρετικά δύσκολες. Θα πρέπει κανείς να κάνει συγκρίσεις μεταξύ συγκρισίμων ε, μέτρων και ε, ειδών. Εδώ δεν είναι η περίπτωσή μας. Τέλος, για να μπορεί κανείς να ε, μετρήσει τις περιόδους απόσβεσης θα πρέπει να λάβει υπόψη του, ε, υπόψη του τις ενεργειακές ε, συγγνώμη, το κόστος της ενέργειας ε, που έχουν ε, υποστεί σημαντικότατες διακυμάνσεις. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, στις χώρες. Έχουμε πολλές περιφέρειες στις 27 χώρες και επομένως το σημείο εκκίνησης του κόστους της ενέργειας είναι τελείως διαφορετικό από χώρα σε χώρα, από περιφέρεια σε περιφέρεια. Υπάρχει και ένα άλλο αμφιλεγόμενο σημείο. Εμείς θέλουμε την εκβάθρον ανακαίνιση. Θέλουμε να χρησιμοποιηθούν τα χρήματα όχι απαραίτητα για ε, πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει και ο ιδιωτικός τομέας και με ε, μικρό χρόνο απόσβεσης. Εμείς θέλουμε εκβάθρον ανακαίνιση, να μην χρειαστεί να επανέλθουμε στα ίδια θέματα μετά από 5 ή 10 χρόνια και είπαμε ότι ανάλογα με το βαθμό ανακαίνηση μπορεί από τα 5 χρόνια να περάσει κανείς στα 10 ή στα 15 χρόνια και παρόλα αυτά ακόμα να είναι συμφέρουσα η διαδικασία. Όσον αφορά τώρα τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, πιστεύουμε ότι οι περισσότερες από τις συστάσεις αυτές είναι σοφές και χρήσιμες και θα προσπαθήσουμε να τι αντιμετωπίσουμε στο νέο κανονισμό. Η προσπάθεια αυτή βασίζεται ε, σε τρία σκέλη. Το πρώτο είναι οικονομικό όπως ξέρετε, η Κομισιόν έβαλε στο τραπέζι την απέτηση για 20% των ε, ε, ε, χρημάτων στις πιο προχωρημένες περιφέρειες και χώρες να αφορούν συγκεκριμένα προγράμματα χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενέργειας στα πλαίσια της προσπάθειας να επιτευχθούν οι στόχοι της στρατηγικής 2020 και βεβαίως και της μείωσης ε, των ε, ε, ρήπων μέχρι το 2050. και 6% να είναι το ποσοστό για τις λιγότερο αναπτυγμένες περιφέρειες. Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο, για πρώτη φορά καθορίσαμε όρους λέμε στα κράτη-μέλη ότι πρέπει να συμμορφώνεστε προς τις απαιτήσει της ε, οδηγίας ε, για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να κάνουν ενεργειακούς ελέγχους, energy audits. Αυτό είναι καινούριο. Δεν υπήρχε όταν υπευλήθησαν και ξεκίνησε η υλοποίηση αυτών των projects. Επίσης έχουμε και τον, τους όρους που απορρέουν από την οδηγία για τα κτίρια. Ε, πλέον υπάρχουν οι όροι αυτοί και αναφέρονται ρητά. Και σε αντίθετη περίπτωση δεν θα δοθούν ε, τα κονδύλια. Επίσης, Πιστεύουμε ότι έχει ευθυγραμμιστεί η ενεργειακή πολιτική μας προς ε, τα, τις συστάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου. Έχουμε δείκτες ας πούμε. Προτείνουμε τρεις ε, δείκτες. Έναν για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Αλλά έχουμε αναθεωρήσει και την μεθοδολογία κόστους-οφέλους και μάλιστα αύριο ε, θα έχουμε και ένα από τα νέα προσχέδια αυτής της μεθοδολογίας και το ελεγκτικό συνέδριο έχει κληθεί να, να ε, συνεκτιμήσει αυτό το προσχέδιο. Θέλουμε και τομιακές προσεγγίσεις ε, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη τους προσεπίτευξης στόχους. Τέλος προωθούμε ιδιαιτέρως τα ε, δημοσιονομικά εργαλεία και την, ε, τα, εργαλεία αυτά της ε, τα οικονομικά τα οποία μπορούν να μας οδηγήσουν σε καλά αποτελέσματα. Έχουμε δει άλλωστε κάποια πρώτα καλά αποτελέσματα στην Λιθουανία. Όπως είπα και στην αρχή πάντως και το ξαναλέω και τώρα, θεωρώ ότι πολλές ιδέες μπορεί να αντλήσει κανείς από την πολύ ε, σωστή και χρήσιμη έκθεση του ε, ελεγκτικού συνεδρίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λανταμπάσο, λέει ο Πρόεδρος. Σχόλια ή παρατηρήσεις επί του σημείου αυτού. Ζωάν Πιέροντι, παρακαλώ. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Να συγχαρώ καταρχάς τους ε, δύο μιλητές για τις πληροφορίες που μας έδωσαν και να του ευχαριστήσω. Η ενεργειακή απόδοση των κτίριων είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν ασχολείται μόνο με τα δημόσια κτίρια αυτή η έκθεση και καλά θα ήταν να το πούμε. Στα δημόσια κτίρια, δεν λέω ότι είναι εύκολο, αλλά είναι πιο εύκολο από τα ιδιωτικά κίνητα στα δημόσια κτίρια λαμβάνονται αποφάσεις από τους άρχοντες που έχουν ε, μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση θα έλεγα σε θέματα ενεργειακής απόδοσης και δεν ενδιαφέρονται τόσο για την ε, αποδοτικότητα την οικονομική. Όταν λοιπόν ε, μιλήσουμε για τον ιδιωτικό τομέα, ευστώ την προσοχή ότι πολλές φορές ε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις ιδιωτικές επενδύσεις και να μην δυσκολεύουμε τα πράγματα. Στην Γαλλία όταν ε, πρόκειται να γίνουν εκλογές υπάρχουν ε, πραγματικά κάποιες διατάξεις άδειε δόμηση που μπορούν να σε τρομάξουν. Καθυστερούν πάρα πολύ δε τις ιδιωτικές επενδύσεις. Θα πρέπει λοιπόν να απλουστεύσουμε τα πράγματα. Θα πρέπει αφενός να δούμε τι γίνεται με τη ρύθμιση και αφετέρου πώς μπορούμε να προωθήσουμε τις επενδύσεις για στον ιδιωτικό τομέα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο θέμα. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπαλσίτης, ο εισηγητής. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση. Κανένας από τους δύο μιλητές, ούτε και εγώ βέβαια, δεν αναφέραμε τη σημασία των δημοσίων συμβάσεων. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στις μείζονες απαιτήσει. Ε, μιλώ δηλαδή για την επιλεξιμότητα, για τη διαφάνεια, τις τιμές κτλ. Οι συνάδελφοί μου φαντάζομαι ότι όλοι θα συμφωνούν ως προς το ότι οι δημόσιες συμβάσεις θα πρέπει να παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην επιλογή των σχεδίων σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση αλλά και σε σχέση και με άλλους στόχους. Ευχαριστώ. Äh, äh, ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο, κύριε Μανκρέβερ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια σύντομη παρατήρηση όσον αφορά αυτό που είπε μόλις ο εισηγητής. Εμείς ακριβώς αυτό κάναμε, δηλαδή ελέγξαμε τις διάφορες διαδικασίες και τις δημόσιες συμβάσεις και το συμβατικό δίκαιο και σκοπός, αν θέλετε, είναι να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι το λιγότερο δαπανηρό και το πιο αποτελεσματικό. Τώρα, όσον αφορά τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί πραγματικά με πολύ θετικό τρόπο αντιμετωπίσατε τις συστάσεις και τις προτάσεις μας. Όσον αφορά τώρα το μέλλον, είμαστε αισιόδοξοι και θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατευθύνεται προς σωστή κατεύθυνση. θεωρούμε ότι οι οδηγίες με αυτόν τον τρόπο μπορούν ευκολότερα να επιτύχουν τους στόχους τους. Μια ακόμα σύντομη παρατήρηση, το ελεγκτικό συνέδριο, όπως είπατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί μια ολοκληρωμένη πολιτική. Βεβαίως και δεν έχουμε τίποτα να πούμε γι' αυτό ότι γίνεται μια αξιολόγηση ενός συνόλου προγραμμάτων. Το θέμα είναι ότι ο στόχος για το 2020, τον οποίο αναφέραμε, 20% μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, είναι πολιτικός στόχος. 17 δισεκατομμύρια έχουμε στη διάθεσή μας. Αυτά τα 17 δισεκατομμύρια θα πρέπει κατά 80 ή 90% να διατεθούν για μέτρα εξοικονόμησης της ενέργειας και καλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας. Και αν κατευθυνθούμε προς αυτό, θα πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε έτσι ώστε αυτό να γίνει σε έναν, με έναν ευχάριστο και αποτελεσματικό τρόπο. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Το ερώτημα του αν οι στόχοι που έχουμε θέσει μπορεί να επιτευχθούν. Είναι ένα γενικότερο ερώτημα, δεν αφορά μόνο την ενεργειακή απόδοση και αν τα μέσα που διαθέτουμε, αν τα μέσα που διατίθενται πραγματικά για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι αρκετά. Γιατί πραγματικά η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 περιλαμβάνει και άλλους στόχους Παραδείγματο χάρη τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων. Το ερώτημα λοιπόν είναι, και βεβαίως αυτό δεν αφορά μόνο εμάς εδώ, αν είναι καλύτερο να ανακαινιστούν κάποια παλιά κτίρια σε κάποιες περιφέρειες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ή το θέμα της ενεργειακής απόδοσης ή το θέμα της βελτίωσης της αγοράς απασχόλησης. Τα μέσα που διαθέτουμε για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και η πολιτική, αν θέλετε, ιεράρχηση αυτών των στόχων. Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για τις τοποθετήσεις σας. Κύριε Μπαλσίτης, θέλετε να ολοκληρώσετε με κάποια επιπλέον σχόλια. Δύο λόγια μόνο κύριε Πρόεδρε. Κάναμε την ανταλλαγή απόψεων. Και είναι φυσιολογικό που θεωρείται σημαντικό αυτό το ζήτημα. Για τις ε, δημόσιες προμήθειες, τους διαγωνισμούς φυσικά και πρέπει να είναι ηλεκτρονικές οι προμήθειες για να εξαλειφθεί, αν θέλετε, η παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Δεν είναι όμως εύκολο αυτό. Και μιλώ τώρα για την επίτευξη των στόχων του 2020. Ακούσαμε τους εκπροσώπους του Ελεκτικού και της Κομισιόν. Ο στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που λειτουργεί στην πράξη και χάρη στο οποίο θα μπορούμε να επαληθεύουμε το αν όλα λειτουργούν όπως πρέπει. Ευχαριστώ. Äh, Σας ευχαριστώ. Τελειώσαμε και με αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξη και το επόμενο θα το συζητήσουμε το απόγευμα. Στις 3 η ώρα θα συνεχίσουμε με την κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ με θέμα η οδηγία ΠΙΦ. Η κυρία Γκερέσλε και ο κύριος Λόπες Αγγιλάρ θα παρουσιάσουν την έκθεσή τους και κατόπιν θα ακούσουμε τον Επίτροπο Σέμετα για την οδηγία PIF.